Bene, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto. Αγαπητοί συναδελφοί, παρακαλώ καθίστε για να αρχίσει η συνεδρίασή μας. Και πάλι με καθυστέρηση. Πρώτο σημείο ημερήσια διάταξη. Την έγκρισή της. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επιφυλάξεις, θα θεωρήσω ότι εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη. Πρώτο σημείο της σημερινή ακρόασης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας που όπως ξέρετε ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου. και είναι τιμή και μεγάλη μου ευχαρίστηση που υποδέχομαι εδώ πρώτο τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών και πρώην Πρωθυπουργό μια τόσο υψηλού επίπεδου παρουσία θα υπάρξει συνέχεια που όλοι ελπίζουμε και ξέρουμε για το πνεύμα αγαστής συνεργασίας που εξέφρασε ο Υπουργός σε όλες τις θέσεις που μέχρι τώρα κατέλαβε. και στο γεύμα εργασίας το οποίο προηγήθηκε της συνεδριασής μας. Και εκεί το ίδιο πνεύμα. Όλοι απάμε εμπειρία γνωρίζουμε ότι συχνά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν είναι οι προθέσεις και τα προγράμματά μας που συγκλίνουν στους στόχους, προς τους στόχους, συνήθως είναι η επικαιρότητα που μας υποχρεώνει να αλλάζουμε κατεύθυνση μερικές φορές. Πάμε χάρη περίπτωση του Ιράν. Δεν προβλεπότανε όπως εξελίχθηκε αλλά όπως είπε ο υπουργό του συναδέλφους μου στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Στοκχόλμη η Σουηδική Προεδρία ενδιαφέρεται πιο πολύ για ορισμένα θέματα. Σήμερα αυτά θα μας τα αναπτύξει ο υπουργό όπως η εταιρική σχέση με τους γείτονές μας προς την Ανατολική Ευρώπη, η στρατηγική για τη Βαλτική, μέσα στα πλαίσια φυσικά των σχέσεων μας με τη Ρωσία. Η διεύρυνση της Ένωσης όταν θα κλείσουν οι συμφωνίες, οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία και τέλος ο πρωταγωνιστικός ρόλος στη διεθνή σκηνή της Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι όσον αφορά την ανάπτυξη. Ένα σωρό προκλήσεις ο χρόνος μικρός και ένα εξελισσόμενο θεσμικό πλαίσιο. Όπως ξέρετε η προσεχής κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας θα επιφέρει και νέες αλλαγές στον τρόπο θεσμικής δράσης μας. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, χωρίς άλλη καθυστέρηση, σας δίνω το λόγο με μεγάλη ευχαρίστηση που θα σας ακούσουμε και που είστε σήμερα παρόν εδώ. Thank you, Chairman. It is an honor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά τα οποία είπατε, αν και κάποια στιγμή άκουγα φινλανδικά. Καλά ακούγονταν, αλλά έχουμε ούτως ή άλλως ε, συναντηθεί και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να πω κάποια πράγματα, λίγα, για να υπάρχει και χρόνος για την συζήτηση που νομίζω ότι είναι το βασικότερο σε ένα κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα με το προφανές θα ήθελα να ξεκινήσω. Ο κόσμος σήμερα είναι πιο απαιτητικός, πιο δύσκολος και πιο επικίνδυνος θα έλεγα από ότι πριν από λίγα μόλις χρόνια είμαστε στην σημεία οικονομικής κρίσης που εμφανίζεται μία φορά ανά γενιά. Οι τελευταίοι αριθμοί της Παγκόσμιας Τράπεζας μιλάνε για απώλεια της παγκόσμιας οικονομίας κατά 3%, μείωση του εμπορίου κατά 10% και από πλευράς εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας τα νούμερα αυτά θα αρχίσουν να έχουν αποτελέσματα στις ασθενείς οικονομίες και τα έθραυστα κράτη και θα έχουν πολιτικές συνέπειες και εμείς θα κληθούμε να βοηθήσουμε για να προσφέρουμε την σταθερότητα η οποία θα κινδυνεύει με ό,τι σημαίνει αυτό. Εάν δείτε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ιστοσελίδα τους έχουν ένα χάρτη όπου φαίνεται πού είναι έτοιμο να παρέμβει και πού έχει παρέμβει τους τελευταίους μήνες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και είναι σαφές το μήνυμα για τους Ευρωπαίους. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προσπαθήσει να δώσει και σταθερότητα στις έθραυστες χώρες και οικονομίες στη γειτονιά μας. Εάν αποτύχουμε σε αυτό θα αποτύχουμε και σε άλλα πράγματα. Ταυτόχρονα, εάν το οικονομικό θέμα είναι, εμφανίζεται μία φορά μόνο κάθε γενιά. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής επίσης είναι κάτι εξίσου σπάνιο. Εντάξει, οι λεπτομέρειες διαφέρουν, αλλά υπάρχει ευρεία συνένεση για την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Για το τι πρέπει να γίνει και για το ότι το ρολόι τρέχει. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αναλάβει τον παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στην πράσινη διπλωματία που είναι απαραίτητη για να ηγηθούμε όλου του πλανήτη στην Κόπενχάγη το Δεκέμβριο για να έχουμε μια συμφωνία για το κλίμα, μια από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτά θα ήθελα να προσθέσω το ότι βεβαίως αυξάνονται οι εντάσεις ε, σε ολόκληρη την περιοχή από την Παλαιστίνη ως το Παντζάμπ και υπάρχουν και στις τεράστιες περιοχές ανατολικά της ε, Ένωσής μας σημάδια γεωπολιτικής γεννητικότητας. 20 χρόνια μετά την ε, κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος, τα οποία θα γιορτάσουμε βεβαίω αυτό το φθινόπορο, μην ξεχνάμε 19 Αυγούστου άνοιξαν τα σύνορα μεταξύ Αυστρίας ε, και Ουγγαρίας ε, και μετά ακολούθησε το Βερολίνο, Πράγα. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τις εκλογές στην Πολωνία μεταμόρφωσαν την Ευρώπη και όλα όσα ακολούθησαν ήταν πολύ σημαντικά. Καταφέραμε να μεταμορφώσουμε την Ευρώπη από ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον πλανήτη σε έναν από τους σημαντικότερους εταίρους για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παγκόσμιας σκηνής τα τελευταία αυτά 20 χρόνια. Αυτό ήταν δική μας επιτυχία. Με τη διεύρυνση, με το ευρώ, με την μεταρρυθμισή των θεσμικών οργάνων. Αλλά εξπακούεται πως όταν έχουμε μεγαλύτερες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, αυτό είναι πρόκληση και για εμάς τους ίδιους και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο, να συνεισφέρουμε να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την αξιοπιστία που έχουμε διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως σε αυτή την περίοδο η Σουηδία αναλαμβάνει για κάποιους μήνες που θα περάσουν γρήγορα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον έχουμε και μια δική μας μεταβατική περίοδο, έχουμε ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έρχεται και η νέα Κομισιόν και ελπίζουμε να κυρωθεί και η σύμβαση της Λισαβόνας κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και μετά άμεσα θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο που λειτουργούν τα θεσμικά όργανα. Όλες αυτές οι κρίσεις, η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εσωτερικές μας αλλαγές είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν από κοινού στους μήνες που έρχονται. Όπως σας είπα μετά από αυτά τα οποία ανέφερα, θεωρώ πως η αξιοπιστία της Ένωσής μας εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα κοντινά σε εμά. Μπορούμε να κάνουμε κηρύγματα για το τι γίνεται αλλού στον κόσμο, αλλά αν δεν αντιμετωπίζουμε τα δικά μας προβλήματα, η αξιοπιστία μας βεβαίως θα έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα. Αυτό ισχύει και όσον αφορά την σημαντική και τώρα πιο υποσχόμενη υπερατλαντική σχέση Πρέπει να δουλέψουμε χέρι με χέρι με τους Αμερικανούς ε, εταίρους μας και με το να δείξουμε και σε αυτούς ότι είμαστε επιτυχείς στην δική μας πλευρά του κόσμου, γινόμαστε και πιο αξιόπιστος εταίρους. Τα άμεσα καθήκοντά μας αφορούν την διεύρυνση και την άμεση γειτονιά μας. Ήμασταν πολύ επιτυχείς και δεν πρέπει να υποτιμάμε το πόσο μεταμορφώνει η έννοια της διεύρυνσης πάρα πολλούς τομείς και πάρα πολλές περιοχές της δικής μας γωνιάς της Ιφιλίου. Υπάρχουν γύρω στα 100 εκατομμύρια άτομα, αν θέλετε, που περιμένουν έξω από την πόρτα μας όταν μιλάμε για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από τους βάρβαρους ε, πολέμους ε, των ε, Βαλκανίων που σημάδεψαν μια δεκαετία της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Σερβία προχωράει προς μια ευρωπαϊκή πορεία, το Κοσμοπέδιο είναι ανεξάρτητη χώρα, στη Βοσνία οι πολιτικοί αντιμάχονται όπως συνηθίζουν οι πολιτικοί, αλλά δεν έχει υπάρξει κρούσμα εθνοτικής βίας στη Βοσνία από όταν τελείωσε ο πόλεμος. Η Κροατία σημειώνει σημαντική πρόοδο της ε, διαπραγματεύσης ένταξης, το Μαυροβούνιο υπέβαλε την αίτηση ένταξης, την προωθήσαμε στο Συμβούλιο, η Αλβανία επίσης υπέβαλε την αίτηση. Για πρώτη φορά λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό, θα έλεγα πως ε, οι δυνάμεις της ε, σύνθεσης στην περιοχή αυτή είναι ισχυρότερες από τις δυνάμεις της αποσύνθεσης της διάλυσης. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε εμεί σε αυτή την περιοχή και το να το κάνουμε νομίζω αποτελεί το βασικό καθήκον μας για τους επόμενους μήνες. Η ευχή μου είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο επίπεδο όσον αφορά τις προοπτικές ένταξης όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Βεβαίως μέχρι να γίνουν μέλη θα περάσει πολύ καιρό για κάποιες από αυτές τις χώρες πρέπει να οικοδομηθούν κράτη εκεί που υπήρχε η Γιουγκοσλαβία και οπωσδήποτε αυτή η δικασία δεν έχει τελειώσει, αλλά υπάρχουν σημαντικά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Εάν όλες οι χώρες κατά τη διάρκεια των επομένων ετών φτάσουν στο ξεκίνημα της διαδικασίας ένταξης με το να υποβάλουν αίτηση με το να περάσουν στη διαδικασία γνωμοδότησης της Κομισιόν, με το να αναπτύξουμε εμείς πολύ πιο φιλόδοξα και πράγματι παρεμβατικά σχέδια μεταρρυθμίσεων για την περιοχή. Θα τους δώσουμε νομίζω μια προοπτική η οποία θα είναι ισχυρότερη από αυτή την οποία έχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν επίσης κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Δεν χρειάζεται να σας τα αναφέρω. Πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση στην ε, Βοσνία να σταματήσουν να κοιτάνε προς το παρελθόν, να στραφούν προς τις Βρυξέλλες και προς το μέλλον, το ίδιο και στην Σερβία. Όλα αυτά γίνονται όμως εάν υπάρχει πολιτική βούληση και όλα αυτά είναι απαραίτητα εάν πρόκειται να διατηρηθεί αυτή η ορμή που υπάρχει σε αυτό το σημαντικό τμήμα της Ευρώπης. Επίσης το ζήτημα της Τουρκίας είναι κάπως επίμαχο και είναι φυσικό αυτό, είναι μεγάλο το ζήτημα, αλλά βεβαίως καθήκον της Προεδρίας είναι να εκτελέσει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις πολιτικές που αποφασίζει η Ένωση και υποστηρίζει και η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Και αυτή η διαδικασία ένταξη πρέπει να προχωρήσει τους μήνες που έρχονται. Ίσως η πιο σημαντική διαδικασία στην Ευρώπη τους ερχόμενους μήνες θα είναι το τι θα συμβεί στην διχασμένη Κύπρο, όπου οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων, ο πρόεδρος Χριστιόφιας και ο κύριος Ταλάτ, έχουν καθίσει και προσπαθούν να ξεπεράσουν, 20 χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, να ξεπεράσουν τον διχασμό της δικής τους πρωτεύουσα και του νησιού τους. Και με το να το κάνουν αυτό, πραγματικά επιδεικνύουν το τι είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν παγιώνει τις διαιρέσεις του παρελθόντος, αλλά τις ξεπερνά και με το να επιδεικνύουν ότι μπορούν να ενωθούν στην Κύπρο θα επιδείξουν πραγματικά ευρωπαϊκό πνεύμα που θα είναι σημαντικό για ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και βεβαίως θα έχει ευρύτερη στρατηγική σημασία για την ενίσχυση της ε, αξιοπιστίας της ευρωπαϊκής διαδικασίας συμφιλίωσης. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους Ένωση ξεκίνησε δύο έργα τεράστιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής σημασίας. Το πρώτο ήταν η, Ένωση, η Μεσογειακή Ένωση πριν από ένα έτος στο Παρίσι όπου αποφασίσαμε να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι σε επαφές μας με τις χώρες της Νοτίας Μεσογείου. Ήδη υπήρχε εδώ και 10 χρόνια η διαδικασία της Βαρκελόνης, αλλά θέλαμε να προχωρήσουμε παραπέρα και αυτό βασίζεται σε απλούς υπολογισμούς. Εάν δούμε τα δημογραφικά στοιχεία αυτών χωρών τα επόμενα 15-20 χρόνια θα αυξηθούν κατά 100 εκατομμύρια στον χώρο τον πληθυσμό τους γύρω σε ένας πληθυσμός δύο φορές ε, η Αίγυπτος. Και άρα είναι σημαντικό το μέλλον τους και για αυτούς και για εμάς. Θα είναι κοινωνίες στάσιμες, απελπισμένες που δεν μπορούν να προσφέρουν δουλειές και δυνατότητες στους πληθυσμούς τους που θα αυξάνονται ή θα είναι κοινωνίες ανοιχτές και οικονομίες ανοιχτές που θα έχουν προοπτικές και αισιοδοξία για το μέλλον, κάτι το οποίο θα έχει τεράστιες επιπτώσεις και για αυτούς και για εμάς. Η Μεσογειακή Ένωση λοιπόν είναι η ουσία της πιο αποτελεσματικής συνεργασίας μας για να τους βοηθήσουμε στην διαδικασία μεταμορφωσής τους που είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Κατόπιν μετά από τη Μεσογειακή Ένωση. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε βεβαίως ε, και τους μετασυσμούς ε, του πολέμου της Γάζας. Έχουμε και την εταιρική σχέση με τις χώρες ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την Κίνα έχουμε 12 διαφορετικές χώρες, έχουμε τα 100 εκατομμύρια της Ανατολικής εταιρικής Σχέσης, έχουμε τα 140 εκατομμύρια της Ρωσίας, τα 60 εκατομμύρια που κατοικούν στην Κεντρική Ασία και με κατέπληξε μια έκθεση που έλαβα πριν από λίγες μέρες και ίσως την έχετε λάβει και εσείς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων που εξετάζει τις σχέσεις μας εκεί πέρα και περιέγραψαν την κατάσταση σε ολόκληρη αυτή την περιοχή με μάλλον άσχημους όρους. Λένε ως εξή. Η πολιτική εκεί είναι ένα τοξικό μείγμα καθυστερημένης δημοκρατίας και αυταρχισμού και βεβαίω συνεχίζει να υπάρχει ο φόβος βίων, συγκρούσεων και τη οικονομικής κρίσης που θα καταστρέψει την περιοχή. Κάπως υπερβολικό ίσως, αλλά όχι εντελώς αναλυθέ. Και πάλι και εκεί πέρα μας ενδιαφέρουν τα πράγματα τα οποία θα συμβούν. Πρέπει η ανατολική εταιρική σχέση να μεταμορφωθεί σε κάτι το οποίο θα είναι σημαντικό για αυτέ τι χώρε που πραγματικά θα εκδιπλώσει αυτές τις δυνάμεις Τη μεταμόρφωσης που έχουμε εμεί και θα τους δώσει ελπίδα για το μέλλον. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με την ε, Ρωσία καθώς οι σχέσεις μας επιδεινώθηκαν πέρσι λόγω της κρίσης με την ε, Γεωργία και τα όσα ακολούθησαν τον συγκεκριμένο πόλεμο, αλλά βεβαίως αλήθεια είναι πως ε, έχουμε συμφέρον να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε την Ρωσία σε μια παγκόσμια και ευρωπαϊκή τάξη που θα βασίζεται σε κανόνες και δεν θα πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας να τους πείσουμε πως τίποτα δεν θα προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στη Ρωσία από την σχέση με όλους τους γείτονές της, ακόμη και τους, τους μικρότερους που βασίζεται σε πραγματική εμπιστοσύνη και φιλία. Έτσι κάνουμε στην Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη. Και για να ολοκληρώσω την εικόνα που σας ζωγράφισα για την Ευρώπη και την άμεση γειτονιά μας, έχουμε μια νέα βόρεια διάσταση αν θέλετε, υπό την έννοια ότι θα πάω στην Στοκχόλμη μεθαύριο και θα δεχτώ την αίτηση της Ισλανδίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αίτηση βεβαίω θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως η αίτηση κάθε άλλη χώρα, λαμβάνοντα βεβαίω πάντα υπόψη πω ε, είναι μέλος της ε, ΕΖΕΣ της, ε, της ζώνης Σέγγεν Οπότε είναι ήδη πολύ προχωρημένη όσον αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οπότε θα συζητήσουμε το μέλλον. Απλά να σημειώσω πως εάν ε, ενταχθεί αυτή η χώρα, θα έχουμε εντάξει μια χώρα που έχει μεγάλη δημοκρατική παράδοση, έχει ένα κοινοβούλιο εδώ και χίλια χρόνια, λίγοι μπορούν να το πούν αυτό και νομίζω θα εμπλακούμε πολύ πιο άμεσα στα στρατηγικά πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα της Αρκτικής. Έχουμε περιβαλλοντικές προκλήσεις, έχουμε δυνατότητες ενεργειακές που είναι ενδιαφέρουσες και η πιθανή και υπάρχουν και βεβαίω οι νέοι πιθανοί διάβλοι που πιθανώ θα ανοίξουν στο μέλλον μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού. Οπότε έχουμε ως Ευρωπαίοι αρκετά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη και στην άμεση γειτονιά μας και βεβαίως θα ενισχύσει την αξιοπιστία μας το να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και στον ευρύτερο κόσμο. Και σε αυτά πρέπει να προσθεθεί πώς αντιμετωπίζουμε και άλλα πολλά ζητήματα από την Παλαιστίνη μέχρι το Παντζάμπ. Πρέπει να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Πριν από ένα χρόνο είχαμε την ε, συνεννόηση Ισραήλ ε, με την ε, Συρία, με επιδιαιτησία των Τούρκων, είχαμε την διαδικασία της Ανάπολης. Ε, υπήρχαν λοιπόν αρκετές διαδικασίες, αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Πρέπει να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα για να μην καταλήξουμε σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση στην Ανατολή από ότι ε, αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε αν μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερότητα του Ιράκ και αν θα αποτελέσει τμήμα των Αμερικανικών και λοιπόν συμμαχικών δυνάμεων, να δούμε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το Ιράν, με το τι συμβαίνει στους ε, δρόμους, ε, όπως έχουμε κάνει τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, και να δούμε αν υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βρούμε μια συνεννόηση στα σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων, αλλά όχι μόνο αυτό, το θέμα των πυρηνικών. Να δούμε επίσης τις εκλογές του Αφγανιστάν και την μετάβαση σε μια νέα φάση ανάπτυξης αυτής της συγκεκριμένης χώρας. Μια νέα σχέση επίσης με το Πακιστάν. Να βοηθήσουμε και αυτή τη χώρα να αντιμετωπίσει και την ασφάλεια και τις οικονομικές και τις λοιπές προκλήσεις που είναι πολύ σοβαρές και να μην ξεχνάμε πως το Πακιστάν είναι σημαντική χώρα. Στο προσεχές μέλλον θα υπάρχουν 200 εκατομμύρια Πακιστανοί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όλα αυτά κατά την άποψή μου συνδέονται και με το τεράστιο ζήτημα της ε, συνολικής μας σχέσης με τον μουσουλμανικό κόσμο. Οι άμεσοι γειτονές μας όχι μόνο στο χάρτη αλλά και στον ίδιο μας το δρόμο στις χώρες μας. Θεωρώ πως υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε μια πιο θετική σχέση. Η Αμερικανική πολιτική άλλαξε. Η σημασία της ομιλίας του Προέδρου Ομπάμα στο Κάιρο δεν πρέπει να υποτιμηθεί. θεωρώ λοιπόν πως η πολιτική τους δεν ε, Βλέπουμε το τι γίνεται Βλέπετε τι γίνεται στο Ιράν με τις εκλογές, το τι γίνεται οπουδήποτε όταν βγαίνει ο κόσμος και διαδηλώνει στην ε, Ινδονησία και αλλού. Δεν είναι οι φονταμενταλιστέ και οι άνθρωποι που δεν έχουν ανεκτικότητα που επικρατούν. Υπάρχουν, όπως υπάρχουν και στις δικές μας κοινωνίες, κάποιες δυνάμεις που έχουν τέτοιε απόψει, αλλά πουθενά δεν πλησιάζουν στο να κυριαρχήσουν. Είναι περιθωριοποιημένοι και άλλες φωνές γίνονται πιο σημαντικές και αυτό κατά την άποψή μου δημιουργεί καλύτερες πιθανότητες για να χειριστούμε τα ζητήματα της ειρήνευσης Μέσης Ανατολής, να σταθεροποιήσουμε το Πακιστάν, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία στο Πακιστάν και να υπάρξει μια συμφιλίωση κάποια στιγμή, ελπίζω, με το έθνος του Ιράν. Το καθεστώς είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν όλες τις χώρες μας, το Κοινοβούλιο και την Προεδρία. Ήταν έντονη η αρχή, έτσι πρέπει να είναι. Ήμουν κάποιες μέρες στα Βαλκάνια, προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα. Μόλις επέστρεψα μετά από τετραήμερη επίσκεψη στο Νότιο Κάφκασο. Πάω στο Κόλμη για λίγες ώρες και μετά ξανά αλλού θα βρεθώ πριν επιστρέψω στις Βρυξέλλες για την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Δευτέρα και βεβαίως για επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως δεν έλυσα με αυτές τις παρατηρήσεις όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε, οπότε περιμένω τις ερωτήσεις σας, οποίες θα προσπαθήσω να απαντήσω και να πω αυτό που, να επαναλάβω αυτό που έχω πει στο παρελθόν η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, επικοδομητικό και νομίζω και αναζωογονητικό για όλους μας και την αναμένω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Η παρουσίαση ήταν και σκέλητη και πλήρης. Εύχομαι και οι συνάδελφοι να μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο. Να σας δώσω ένα, μια σημαντική πληροφορία οργανωτική για σήμερα. Ο Υπουργός θα φύγει σε μία ώρα και κάτι. Έχω 34, τα ονόματα 34 συναδέλφων που ζήτησαν να μιλήσουν. Σας παρακαλώ λοιπόν τα εξής δύο. Πρώτο, ο κατάλογος των αγοριτών κλείνει αυτή τη στιγμή. Δεχτείτε το. Δεύτερο, δυστυχώς, σας παρακαλώ, δείξτε την ευγένεια να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά κατά άτομο για να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν όλοι. Αρχίζουμε με τους συντονιστές των ομάδων και μετά θα ακολουθήσουμε με τους υπόλοιπους αγορητές. Πρώτος, ο συνάδελφος Σαλαφράνκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε εκ μέρου του συναδέρφου Έλμαρ Μπρόκ αλλά και όλων των συναδέρφων από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλω να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Μπίλτ και να του ευχηθώ καλή τύχη κατά την ε, θητεία του. Και του εύχομαι καλή τύχη γιατί σίγουρα οι προκλήσεις που έχει μπροστά του είναι πολλές και μεγάλες. Το δημοψήφισμα για την επικύρωση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η νέα επιτροπή που μένει να εκλεγεί, οι συνδρίες τη Κοπεχάγη όσον αφορά το πρωτόκολλο του Κιώτο και βέβαια η οικονομική κρίση που είναι πολύ σοβαρή. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, κύριε Προεδρεύοντα, τρει ερωτήσει έχω. Πρώτον, θέλω να σα πω ότι από τη δικιά μα πολιτική ομάδα συμμεριζόμαστε την άποψή σα για μια ισχυρή Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι ετοιμάζει η Σουηδική Προεδρία προκειμένου να διασφαλίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα την θέση σε ισχύ των εξωτερικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα πρέπει να ξέρετε ότι συμμεριζόμαστε την αποψή σα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ότι δηλαδή πρέπει να ισχύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε πολύ συγκεκριμένα θέλω να σας ρωτήσω, μια που αναφερθήκατε και εσείς λίγο στην αρχή, για το Ιράν. Η πρόταση που έκαναν οι μεταρρυθμιστές, ο τέος πρόεδρος Χαταμή για παράδειγμα, για την εισαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος, μια νέα διαδικασία που θα επικυρώσει όχι τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών. Τέλος, για τις Ονδούρες θέλω να μα πείτε λίγο κύριε Προδρεύοντα εδώ. Βλέπετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ασχοληθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εννοείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει τη δημοκρατική ομαλότητα και σταθερότητα στην περιοχή. Ξέρουμε τι έχει κάνει ο πρόεδρος Κωνσταντίνο η ερώτησή μου είναι η εξή. Η Συμφωνία Σύνδεσης, στην οποία καταλήγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, επηρεάζεται από την κατάσταση στις Ονδούρες. Ή, τελειώνω πρόεδρε, ή πιστεύετε ότι την Τετάρτη που είναι η προθεσμία που έχει δώσει ο πρόεδρος της Κωνσταντίνα θα ξέρουμε περισσότερα για να δούμε τι θα κάνουμε με τη Συμφωνία αυτή σύνδεσης. Ευχαριστούμε κύριε Σαπάκα. Σχεδόν σεβαστήκατε το χρόνο των δύο λεπτών. Ο κύριος Φόποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε πάρα πολλά πράγματα, όλα σημαντικά. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα που ετέθη εμέσως στην Ολομέλεια για τα Βαλκάνια. Δύο σύντομα ερωτήματα. Το ένα αφορά τις σχέσεις Κροατίας-Σλοβενίας. Θέλετε κάποια νέα πρωτοβουλία ή θα περιμένετε ή θα εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία της νέας κυβέρνησης ή του νέου πρωθυπουργού στην Κροατία για να ξεκινήσουν ξανά συνομιλίες. Δεύτερον, ζητήματα θεωρήσεων δεν είναι μόνο δική σας ευθύνη. Εγώ δεν είμαι κατά της λύσης που βρέθηκε, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένας ε, τρόπος να ενταχθεί και η Βοσνία σε αυτή την ε, συμφωνία. Βλέπετε να υπάρχει ένας ε, τέτοιος τρόπος και πώς θα μπορέσουμε να τελειώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα με την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Σας ευχαριστώ. Ora la parola l'onorevole Kacin. Ο κύριος Κατσίν. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα, θα συνεχίσω με την Βοσνία Ριζεγοβίνη, γιατί βλέπετε μου έρχονται διάφορα απελπισμένα email τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τις συνέπειες της ανακοίνωσης ε, για την Βοσνία ότι δεν θα στηριχθούν όσον αφορά το καθεστώς της 1ης Ιανουαρίου. Έτσι όπως βλέπουν εκείνοι λοιπόν τη θέση τους, πραγματικά βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση. Θεωρούν τους αυτούς τους θύματα σε μία περίοδο Βαλκανικών πολέμων επίσης είχαν εμπάργο για πολεμικό εξοπλισμό. Τότε ήταν επίσης θύματα λοιπόν και τώρα πάλι είναι θύματα όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Οι Σέρβοι, οι Κροάτες βλέπετε δεν χρειάζονται τίποτα παραπάνω, όμως η Βοσνία χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα κύριε Υπουργέ να τους βοηθήσετε, να φροντίσετε να μπορέσουν να έχουν συγκεκριμένη αρρωγή και βοήθεια όσον αφορά την δίκηση της χώρας τους και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που υπάρχουν για να προδεύσουν και να πετύχουν την ελεύθερη κυκλοφορία των Βοσνίων πριν από το 15η επέτειο της Δεβερνίτσα που είναι του χρόνου. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει και το Πέδιο όσον αφορά δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Αντίθετα όμως έχουν ξεχαστεί. Εγώ λοιπόν πιστεύω κύριε Υπουργέ ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας εσείς θα πρέπει να εξισορροπήσετε κάπως την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Αλλιώς οι συνέπειες θα είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η συνάδελφος Λούνατσεκ έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ναι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, που είσαστε και κεφαλής του Συμβουλίου, εκτιμάω απόλυτα το γεγονός ότι έρχεστε εδώ, παίρνετε λίγο χρόνο να συζητήσετε μαζί μας και το εκτιμάω πραγματικά όλος ιδιαίτερος ότι μας μιλάτε για τις επιθυμίες της Προεδρίας σας, τι θέλει να κάνει και το νιώθουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει ηγετικό ρόλο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πολύ θετικό αυτό. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η καλή ρητορική που μας παρουσιάζεται εδώ σήμερα να βρει ανταπόκριση και στην πράξη. Για παράδειγμα, η ιδέα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου αυτές να έχουν πραγματικά αρκετά χρήματα. Αυτό μερικές χώρες το αρνούνται, άλλες το θέλουν πολύ. Λοιπόν, για το ταμείο αυτό θέλω να ξέρω περισσότερα. Έπειτα, ερωτήσει μου. Όπω είπαν και οι προλαλήσαντε, έτσι και εγώ θέλω να ανηφερθώ λιγάκι στο θέμα των θεωρήσεων ε, και τα Βαλκάνια. Το Μαυρό Βούνιο, η Μακεδονία, η Ομιλήτρια θα έχουν τη διευκόλυνση. Με τη Βοσνία όμω τι θα γίνει. Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Οι τρει τελευταίοι ειδικοί απεσταλμένοι για τη Βοσνία, ο τελευταίο ομιλούσε επέκριναν την Επιτροπή για την πρότασή της, που δεν έχει συμπεριλάβει τους Βόσνιους αυτήν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το Συμβούλιο να κάνει ό,τι χρειάζεται και να βοηθήσει τους Βοσνίους να περάσουν σε αυτό το καθεστώς ελευθέρωσης από τη Βίζα, να μην τους είναι αναγκαία, μέχρι τα τέλη της χρονιάς, ώστε να μπορέσουν να έχουν την ελευθερία όλοι οι Βόσνοι, έτσι όχι μόνο οι Σέρβοι και οι Κροάτες, οι Βόσνοι Βόσνοι να μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα μετά από το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Τέλος θέλω να σε ρωτήσω για το Ιράν. Μέσα Αυγούστου θα έχουμε την αρχή, ας πούμε, της εκλεγμένης εντό αγωγικών ε, του Αχμεντίν Μουνιτζάτ και ελπίζω ότι εσείς και τα κράτη-μέλη δεν θα εκπροσωπηθείτε σε υψηλό επίπεδο στα γένεια της νέας αυτής κυβέρνησης. Γιατί πρόκειται για πάτη. Οπότε εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε. Ευχαριστούμε. Τάνοκ τώρα, για δύο λεπτά παρακαλώ. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, για τη Μέση Ανατολή, για να επανέλθω στην τσεχική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των σχέσεων μας με το Ισραήλ, θα επανέλθει στο πρόγραμμά σας, είναι πιο δύσκολο τώρα με τη νέα κυβέρνηση. Και καθώς υπάρχουν ε, προτάσεις για να ψυχρανθούν η σχέση με το Ισραήλ. Πώς αυτό θα βοηθήσει τους ε, θανάσιμους ε, εχθρούς του Ισραήλ, όπως η Χεσμολάχ, η οποία δραστηριοποιήθηκε, όπως ξέρετε, στο Λίβανο προς ε, έκπληξή μας. Επίσης, για την Ασία δεν αναφέρατε τη Σρι Λάνκα, που βρίσκεται σε μια διαδικασία νοικοδόμησης μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Είχε παίξει σημαντικό ρόλο η Σουηδία στο παρελθόν, αλλά τώρα γεμίζει ένα κενό που υπάρχει εκεί πέρα η Κίνα όσον αφορά την επιρροή. θα επανέλθει η δική μας επιρροή, γιατί η Κομισιόν βεβαίως έχει κακή φήμη, φοβάμαι, στο Κολόμπο τα τελευταία χρόνια. Και Βεβαίω ε, θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειάζονται καλύτερη προσέγγιση. Βεβαίω στην Κύπρο οι διμερεί επαφέ μεταξύ του Προέδρου Χριστόφια και του κ. Ταλάτ είναι πολύ σημαντικέ και υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ, αλλά το, ε, το βεβαίω βρίσκεται στην Άγκυρα και μάλλον στο Υπουργείο Άμυνα και στον τουρκικό στρατό. Έχετε κάποιες ενδείξεις πως η Τουρκία θα αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας που ε, έχει υπογράψει εδώ και δύο-τρία χρόνια. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Τώρα εκ μέρους της ΓΚΟΕ, συνάδελφος Χατζηγεωργίου. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Καλμπίλτ, να τον συγχαρώ για την παρουσία του εδώ, να συγχαρώ και τον Πρόεδρο για την εκλογή του την προηγούμενη συνεδρία. Ε, θα αναφερθώ λίγο στη διεύρυνση, κύριε Μπίλτ, ε, στην οποία αναφερθήκατε και θα πω δύο πράγματα για την Τουρκία και να ρωτήσω κάτι. Στην Κύπρο ασφαλώ σήμερα διεξάγονται συνομιλίε μεταξύ του Προέδρου τη Δημοκρατία του κ. Χριστόφια και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του κ. Ταλάτ. Είπατε ότι μια πιθανή λύση θα είναι μια υπογράμμιση των ευρωπαϊκών αξιών. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι θα αποτελούμε, εάν τα καταφέρουμε στην Κύπρο, γιατί προέρχομαι από την Κύπρο, ένα παγκόσμιο σύμβολο ε, συνένωσης δυνάμεων διαφορετικών κοινοτήτων και ο στόχος μας είναι πολύ ειλικρινά ε, αυτή η λύση να επιτευχθεί. Ε, πάνω απ' όλα εμείς οι Κύπροι είναι που χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη τη λύση να μην ταξιδεύουμε μόνο ελεύθερα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά πρώτα απ' όλα στον ίδιο μας τον τόπο. Όμως καταλαβαίνετε ότι οι δυνατότητες των δύο ηγετών στην Κύπρο είναι να λύσουν πιθανώς εσωτερικές πτυχές του κυπριακού προβλήματος. Δεν μπορούν, υποθέτω, να λύσουν το πρόβλημα της τουρκικής κατοχής. Δεν έχουν αυτή την δυνατότητα ούτε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ε, δεν έχουν την δυνατότητα να, πούν τι θα γίνει στο θέμα των εγγύσεων. Μια ανεξάρτητη Κύπρος ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρειάζεται εγγύησει ξένων κρατών. Στην Κύπρο, κύριε Μπίλτ, σήμερα υπάρχουν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες για 80.000 Τουρκοκύπριους. Ένα στρατιώτης για κάθε δύο πολίτες. Ούτε οι ευρωβουλευτές δεν έχουν τέτοια ασφάλεια την οποία δεν χρειάζονται ασφαλώς οι Τουρκοκύπροι. Είναι μια παρουσία τουρκικού κατοχικού στρατού σε ένα κράτο μέλο. Επανυπογραμμίζω ότι εμεί πρώτοι θα θέλουμε τη λύση, αλλά θέλω να ρωτήσω ποια πίεση μπορεί να ασκηθεί επιτέλου στην Τουρκία για να υλοποιήσει το πρωτόκολλο, να ανοίξει τα λιμάνια της, τα αεροδρόμια της προς την Κύπρο, να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, πράγματα τα οποία θα σπρώξουν προς την λύση. Ε, κλείνω με μια αναφορά στο Παλαιστινιακό, ε, κύριε Μπίρτ. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο συγκεκριμένη στο τι βοήθεια μπορεί να παράσχει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Τώρα με την παρέμβαση του κυρίου Πλεύρη, του κυρίου Πλεύρη, κλείνουμε με τους συντονιστές. Μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Υπουργό. Κύριος Πλεύρης. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ε, ρωτήσω κάποια πράγματα για τη διεύρυνση την οποία αναφέρατε ως προς την πλευρά της Ανατολής. Ε, πώς απαντάτε στα επιχειρήματα των κυβερνήσεων που έχουν τοποθετηθεί της Γαλλίας και της Γερμανίας ότι με την Τουρκία δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ Πλήρη ενταξιακή πορεία αλλά ειδικέ σχέσει, ένα ειδικό καθεστώς και αν τυχόν πιστεύετε στον ευρωπαϊκό ε, προσανατολισμό της Τουρκίας ε, θεωρείτε ότι τα σύνορα της Ευρώπης μπορούν να φτάσουν μέχρι το Ιράν και το Ιράκ αυτομάτως εκεί πέρα δεν ξεφεύγουμε ουσιαστικά από αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, θα ήθελα επιπλέον να τονίσω και εγώ αυτό αναφορικά με την Κύπρο κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να πιεστεί η Τουρκία ώστε να αναγνωρίσει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά για τη μετανάστευση, γιατί δεν άκουσα την τοποθέτηση της, ε, τη δική σας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο κύμα παρανόμων μεταναστών προς την Ευρώπη. Κυρίως ε, οι μεσογειακές χώρες πληρώνουν αυτό το τίμημα. Θεωρείτε ότι από τη δική σας πλευρά, ενώ από την πλευρά των εξωτερικών υποθέσεων μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τις χώρες που στέλνουν μετανάστες να δέχονται την επαναπρόθεση και επανέρχομαι πάλι στο θέμα της Τουρκίας μπορεί, γιατί είναι μια transit χώρα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει την Τουρκία και να την υποχρεώσει να τηρήσει τις ε, συμφωνίες που υπάρχουν για την επαναπρόθεση θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό που είπατε τώρα για το Ιράν ε, θεωρείται ότι μπορούμε να τα βρούμε με το έθνος, αλλά με το καθεστώς τι θα γίνει. Διότι όπως καταλαβαίνετε, ε, για να τα βρούμε με μια χώρα πρέπει να τα βρούμε και με το καθεστώς. Θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν. Και θα ήθελα και εγώ και την τοποθέτησή σας για την Ονδούρα και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση. Ειδικά όμως για το θέμα το μεταναστευτικό θα ήθελα την τοποθέτηση σας. Ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε σεβαστεί μέχρι τώρα το χρόνο μας. Το λόγο στον κύριο Υπουργό, ο οποίος μπορεί να έχει το χρόνο που θέλει. Αλλά αν θέλετε να δώσετε χρόνο και για άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να εξακολουθήσει να είναι λιτός όπως και πριν. Δύο λεπτά φυσικά δεν μου φτάνουν. Παραπάνω, παραπάνω λέει ο Πρόεδρος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο χωρίς να αποφύγω πολλέ ερωτήσει. Για την κύριο Σαλαφράγκα, προετοιμασία για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Καταρχήν, πρέπει να περιμένουμε την κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό που οφείλουμε να κάνουμε αν και όταν κατ' ελπίδα θα κυρωθεί η συνθήκη. Θεωρώ την υπηρεσία αυτή πάρα πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον και πρέπει να λυθούν, επιληθούν καταρχήν ορισμένα θέματα. Πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες αποφάσεις, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι διανοητικά και πολιτικά, να έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά πρέπει όμως να σεβαστούμε την διαδικασία, τη θεσμική που ισχύει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την Ιρλανδία και θα πρέπει να περιμένουμε για λίγο, χωρίς να κοιμόμαστε βέβαια, αν επιτρέπεται η περιγραφή αυτή όσον αφορά την κατάσταση. Ονδούρα. Το συζητήσαμε κάπου σύντομα στην Ολομέγια της προάλλες Νομίζω ότι σας είπα στην Ολομέλεια ότι πιστεύουμε ότι η νέα προσπάθεια του Προέδρου Αρίας το Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο θα είναι επιτυχής. Δεν συνέβη αυτό για το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Και η πολιτική που τώρα ακολουθούμε είναι πάνω κάτω αυτή που σας περιέγραψα την περισμένη εβδομάδα. Πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Μεσολαβή. Αυτή είναι η δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή να επιληθεί η διαφορά αυτή. Όλες οι άλλες εναλλακτικέ λύσει είναι κακέ. Και είμαστε σε άμεσο διάλογο και με αυτόν την οργάνωση των Αμερικανικών κρατών σχετικά με το πώ εμεί ω Ένωση μπορούμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα υποστήριξη των προσπαθειών του Προέδρου Αρία. Και α ελπίσουμε και α προσευχόμαστε ότι θα πετύχει. Αν δεν πετύχει, τι θα κάνουμε στη σχέση μας με τις διαπραγματεύσεις με την Κεντρική Αμερική. Ελπίζω να μην χρειαστεί να φτάσουμε ως εκεί. Ας περιμένουμε αν υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα δούμε τι θα κάνουμε τότε. Προς το παρόν, ποντάρουμε στις μεσολαβαστικέ προσπάθειες. Μερικέ ερωτήσεις για το Ιράν. Φυσικά, προτιμώ να μην πω σε λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή σχετικά με το τι θα έπρεπε να κάνει το Ιράν, με δημοψηφίσματα, τις εκλογές κλπ. Είναι μια χώρα που έχει ένα είδο πολυφωνία μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο πλαίσιο. Και πιστεύω ότι γίνεται συζήτηση μέσα σε αυτό το περιορισμένο πλαίσιο πώ να χειριστούν αυτά τα θέματα. Α δούμε τι θα βγει από τη συζήτηση αυτή, Α περιμένουμε. Αυτοί είναι οι ηγέτε στο Ιράν. Αυτοί οι ηγέτε στο Ιράν θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την νομιμότητα των διαδικασιών στα μάτια αυτών που εκλέγουν. Τώρα, σε τι πορίσματα θα καταλήξουν, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως αυτό θα επηρεάσει την κατάσταση. Εμείς θέλουμε να έχουμε επαφή με το έθνος του Ιράν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έθνος. Έχουμε νέους με ελπίδες, με όνειρα, με προσδοκίες όπως όλοι και να το ισοσταθμίσουμε αυτό με την βιαιότητα που είδαμε στους δρόμους τον τελευταίο καιρό είναι δύσκολο πράγμα. Σχέσεις με το καθεστώς είπατε να έχουμε. Φυσικά έχουμε διπλωματικές σχέσεις. Και συζήτησα με τον Υπουργό Εξωτερικών Μοντάκη κάποιες φορές τις τελευταίες εβδομάδες. Και από τη Βρετανική Πρεσβεία εκεί, όπως ξέρετε, γίνανε ορισμένα επεισόδια. Είχαν προβλήματα, τους ε, είχαν κράτηση, απελευθερώθηκαν τελικά. Ε, μια κοπέλα, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμιά εξήγηση, κρατήθηκε από τις αρχές. Φυσικά έχουμε διάλογο με τις Ιρανικές αρχές σε όλα τα επίπεδα, να απελευθερωθεί και αυτή. Συγκεκριμένα λοιπόν, ναι έχουμε επαφές το ίδιο πράγμα για τα πυρηνικά και για άλλα θέματα. Πρέπει να χειριζόμαστε θέματα σε σχέση με την πραγματικότητα που ισχύει εκεί. Και ας περιμένουμε να δούμε θα, ποια θα είναι η έκβαση όλων αυτών. Προχωρώ. Βαλκάνια, συγκεκριμένα Βοσνία, το θέμα της ε, βίζας. Για την Κροατία και ε, ε, και τη Σλοβενία ε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτό που αναφέρθηκε. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Για την Κροατία και τη Σλοβενία, αυτό που είπα και ιδιωτικά και το λέω και δημόσια τώρα, Νομίζω υπήρξε όξυνση των τόνων και από τι δύο πλευρέ. Στα Βαλκάνια πρέπει να είναι κανεί πολύ προσεκτικό με τα λόγια του. Πολύ προσεκτικό με τα λόγια του. Γιατί υπάρχουν και ορισμένα άτομα που τελικά πιστεύουν αυτά που λένε και αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρέ συνέπειε. Καλό λοιπόν τους ηγέτες και από τις δύο πλευρές να είναι λίγο πιο ήρεμοι, cool down τα λόγια, να τα σκέφτονται πριν τα λένε και οι δυο έχουν συμφέρον να επιληθεί το θέμα αυτό και όσο πιο σύντομα το κάνουν τόσο καλύτερα και για την Κροατία γιατί όλοι έχουμε συμφέρον στο να συνεχιστεί, να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξη τη Κροατία. Είναι σημαντικό και για τη χώρα αυτή και για όλε τι σχέσει μα με την περιοχή αυτή, αλλά είναι σημαντικό και για τη Σλοβενία. Καμία χώρα δεν θέλει να αισθάνεται ότι απομονώθηκε στην Ένωση. Δεν το θέλουμε αυτό ούτε εμεί. Κανένα δεν το θέλει. Λίγο περίοδο περίσκεψη θα του βοηθήσει λοιπόν και αυτού. Γιατί αυτό είναι η Ευρώπη. Να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουμε επικοδομητικά. Και να είμαστε και έτοιμοι για συμβασμούς. Το πρόβλημα της Βοσνίας τον άφεραν οι βουλευτές. Ξέρω τι λέγεται αυτή τη στιγμή, ποιοι είναι οι τόνοι στο Σεράγεβο, αλλά δεν είναι καινούργιο αυτό το πρόβλημα. Το ξέραμε. Και θα έπρεπε και αυτοί να υποψιάζονται ότι θα πάρει τη διάσταση που πήρε. Με τον Καρλ Σφάντσεμπερ, τον Μπερνάρ Κουσνέρ, μια ολόκληρη μέρα εξοδέψαμε να συζητάμε με την Βοσνιακή ηγεσία από όλα τα κόμματα και τους είπαμε πρέπει να συνεργαστείτε. Αν δεν συνεργαστείτε και αν δεν πάρετε τις αναγκαίες αποφάσεις για την απελευθέρωση της βίζα, θα χάσετε το τρένο. Δεν μπορεί να μπλοκάρονται όμοιροι όλα τα, Βασκά, τα Βαλκάνια στους, λόγω των Βόσνιων πολιτικών. Χρειάζεται επιτάχυνση αυτό το τρένο. Τώρα, το κατά πόσον βάρινε αυτό και μέτρινε, βάρινε, αλλά όχι αρκετά. Πήγε και ο Αμερικάνος υπουργό εκεί. Μία μέρα, τα ίδια πράγματα, με την ίδια ηγεσία. Τα ίδια τους έλεγε. Τους είπε, ναι, πρέπει να δράσετε από κοινού. Περισσότερη δράση, πάρτε απόφαση. Βιομετρικά κλπ πρέπει να εξασφαλιστεί αξιοπιστία όχι μόνο με του υπουργού εξωτερικών τη Ευρώπη. Είμαστε, είμαστε καλοί άνθρωποι. Με του υπουργού εσωτερικών και είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Καλοί άνθρωποι είναι και αυτοί, δεν λέω. Αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Πρέπει να πετύχετε αξιοπιστία τη δική σα και με αυτού. Και τα καλά λόγια και οι κατηγορίε κατά τη διεθνή κοινότητα δεν σα βγάζουν πουθενά, δεν σα πάνε πουθενά. Ελπίζω λοιπόν ότι οι Βόσνιοι ηγέτες έχουν αρχίσει να συνεργάζονται για δράση. Είπατε είναι θύματα. Το ξέρω το σύνδρομο αυτό. Μερικές φορές αποκαλώ την Βοσνία δεύτερη πατρίδα μου, γιατί έχω περάσει πολλά χρόνια εκεί. Είναι θύματα της ανικανότητας των πολιτικών ηγετών τους να συμφωνήσουν. Και πολλοί από αυτούς, και το λέω αυτό ομά και ανοιχτά, λένε δώσαμε έναν πόλεμο, κάναμε έναν πόλεμο πριν από 15 χρόνια. ας φροντίσουν για τους νέους τους τι θα γίνει, τι θα κάνουν στην Ευρώπη. Οι νέοι δεν θέλουν τους πολιτικούς που μαλώνουν, θέλουν το ευρωπαϊκό όραμα και οι Βόσνιοι πολιτικοί πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε θέση από κοινού να πάρουν τις αποφάσεις που θα τους βάλουν στην Ευρώπη. Και αν το κάνουν αυτό θα είμαι ο πιο ευτυχής άνθρωπος στον κόσμο. Αν δεν το κάνουν όμως, στην, ε, στην Ένωση δεν μπαίνει κανείς τζάμπα. Χρειάζεται προσπάθεια. Κόσοβο. Χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ λεπτό και αυτό το θέμα. Υπάρχουν και ορισμένα θέματα ενδοευρωπαϊκής νομιμότητας. Χρειάζεται επικοδομητική δράση και νομίζω ότι μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά. Για τα θέματα για το κλίμα. Νομίζω ακούσατε τον Σουηδό Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια της προάλλες. Δεσμεύτηκε ότι θα είναι προτεραιότητα για μας στο εξάμεινο αυτό το θέμα. Και όλοι τον υποστηρίζουμε σε αυτό. Θα υπάρχει πράσινη διπλωματία εκ μέρους της Σουηδίας το εξάμεινο. Αυτό που ρωτήσατε το Ιράν δεν τα απάντησα ούτε τις πράλες, ούτε και σήμερα απαντώ. Δεν διαφωνώ με αυτά που είπατε, δεν διαφωνώ απόλυτα για τον κύριο Τάνοκ. Κάμποσα θέματα. Ισραήλ. Θέλουμε ένα βαθύ διάλογο με το Ισραήλ για το μέλλον, σίγουρα. Και αυτό ισχύει για όλου. Ιδιαίτερα όταν έχουμε διαφωνίε. Έχουμε μερικέ σοβαρέ διαφωνίε αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ. Χρειαζόμαστε διάλογο για να δούμε αν μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε θέματα. Το ίδιο και οι Αμερικάνοι. Είναι σε διάλογο με το Ισραήλ έχει σχέση και με τους ε, επικισμούς, μια συγκεκριμένη πολιτική, αν θέλει κανείς να ασχίσει μια ειρηνευτική πολιτική. Έχουμε το θέμα της Γάζας. Εμείς από τον πόλεμο της Γάζας έχουμε σαφή θέση ότι η απομόνωση δεν είναι και ηθικά απαράδεκτη, αλλά ουσιαστικά δεν αποδίδει. Και για τους Ισραηλινούς δεν αποδίδει ως θέση και ελπίζουμε ο διάλογος με το Ισραήλ να τους κάνει να το δούνε αυτό να χαλαρώσουν την πολιτική που ασκούν. Και μετά από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα αναπτυχθούν οι σχέσεις μας. Πάντως τυπικά βήματα αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να γίνουν. Το Σρι Λάνκα είναι και αυτό ένα θέμα που το παρακολουθούμε. Είχαμε ένα είδος ε, θριαμβολογίας εκ μέρους της ε, κυβέρνηση του Κολόμπο μετά τα πρόσφατα γεγονότα και δεν ήταν έτοιμοι να ακούσουν τι έχει να τους πει η διεθνής κοινότητα. Είχαμε την επίσκεψη του Ιμπάν Κιμούν και τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν να έχουν πρόσβαση στα στρατόπεδα, τους το αρνήθηκαν. Ταυτόχρονα όμως η ηγεσία εκεί βλέπει ότι το να κερδίσει την ειρήνη είναι πολύ πιο, γρήγορα, πιο δύσκολο από το ότι να κερδίσει τον πόλεμο. Είναι εύκολο να κερδίσει τον πόλεμο γιατί η σταθερότητα τη χώρα χρειάζεσαι η ειρήνη. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει το μυαλό και την ψυχή των ανθρώπων και χρειάζονται τη βοήθεια τη διεθνού κοινότητα. Κάποια στιγμή θα είμαστε αναγκαίοι για αυτού και θα μα καλέσουν και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτή τη στιγμή. Κύπρος. Η Ένωση δεν μπορεί να παίξει ρόλο στη διαδικασία που αυτή τη στιγμή κινείται στην Κύπρο. Είναι θέμα για τον πρόεδρο Κριστόφια και τον ε, κύριο Ταλάτ, ηγέτες των δύο κοινοτήτων, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν. Με εντυπωσιάσουν και οι δύο για την... το πιστεύω τους ότι θέλουν να το πετύχουν αυτό. Ούτε η ιστορία, από την ιστορία τους και από το background τους, νομίζω πραγματικά θέλουν να το πετύχουν, αλλά υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες. αλλά δεν είναι πιο σοβαρέ από εμπόδια που έχουμε ξεπεράσει στο παρελθόν σε άλλε περιπτώσεις. Αν ξεπεράσουν το θέμα του governance, της διακυβέρνησης, που είναι πολύ λεπτό, πιστεύω ότι τα άλλα θέματα είναι δυνατόν να επιληθούν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη που στηρίζεται σε άλλες εμπειρίες μου από το παρελθόν. Υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία αναφερθήκατε, ασφάλεια κλπ. Αυτά είναι από τα πιο δύσκολα θέματα και πιστεύω ότι θα πρέπει προς το τέλος να τα συζητήσουν και αυτά. Θα ήταν άτοπο εκ μέρους μου να προσπαθήσω να παίξω κάποιο ρόλο για τα θέματα αυτά. Τονίζω ότι είναι σημαντικά. Και μετά έχουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου, όπως και εσείς και άλλοι επενηχθήκατε και αναφέρατε το εμπόριο, πρωτόκολλο της Άγκυρας, όλα αυτά θα, όλες αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου που έχουμε λάβει θα πρέπει να τις ξαναδούμε κάποια στιγμή να εφαρμόζονται σωστά και από μας και από άλλους. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και αν υπάρξει συμφωνία, πολύ ελπίζουμε να υπάρξει, εμείς τότε ως Ένωση θα είμαστε έτοιμοι να την υποστηρίξουμε, να την αγκαλιάσουμε ας πούμε. Γιατί πιστεύω ότι τα οικονομικά ωφέλη της συμφωνίας θα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τις δύο κοινότητες αυτά τα οικονομικά ωφέλη μπορούν να έρθουν μετά από μερικά χρόνια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε, να βοηθήσουμε τη συμφωνία. Αλλά η επίσκεψη της συμφωνίας δεν είναι δικό μας έργο. Είναι έργο των δύο ε, ανθρώπων που ανάφερα στην Κύπρο. Μετανάστευση. Όντω. δεν είπα τίποτα για τη μετανάστευση και ο λόγος είναι διότι είχα μια επίσημη συνάντηση των άλλων υπουργών, στους οποίους αναφέρθηκα πριν, Υπουργοί Δικαιοσύνη και Εσωτερικών, που είναι υπεύθυνοι για τη μετανάστευση, στη Στοχόλμη τη προάλλε και σα ομολογώ ότι δεν ξέρω τι είπανε. Δεν έχω ιδέα τι είπανε. Εγώ ήμουν στον Νότιο Κάφκασο, δεν ξέρω τι συζήτησαν. Πάντω το θέμα θα είναι στην μίληση διάταξη του Συμβουλίου του Οκτωβρίου με βάση αποφάσει που ε, ε, ελήφθησαν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη από τους συναδέλφους. Θα μου επιτρέψετε να περιορίσω κι άλλο το χρόνο των αγοριτών 1,5 λεπτό maximum. Γιατί έχουμε περίπου άλλους 30 αγορητές. Ο κύριος Μπροκ πρώτος. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα για την περαιτέρω διεύρυνση. Είπατε πως η Ισλανδία θα υποβάλει μεθαύριο την αίτησή της και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι μέρος ήδη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οπότε έχει τυπικά τουλάχιστον ενσωματώσει ένα μεγάλο μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. Σε τι διαφέρει αυτό από τις υπόλοιπες περιπτώσεις της ε, διεύρυνσης. Εσείς ο Σουηδός έχετε εμπειρία από το να ανήκει κανείς στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μήπως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο ενίσχυσης της ε, ανατολικής ε, εταιρική σχέσης. Και να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσει, κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω καθυστερήσει, χωρί να σημαίνει ότι οπωσδήποτε δεν θα γίνει αυτό. Σα ευχαριστώ. Κύριε Ρότσεκ. E Ενάμιση λεπτό πάντα. Ναι, ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα επέβαλε θεωρήσεις στη Τσεχική Δημοκρατία ο Καναδάς. Τι πρέπει να κάνει η Τσεχία μαζί με τη Σουηδική Προεδρία ώστε να αλλάξει την απόφαση αυτή ο Καναδάς και να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση όπου δεν χρειάζονταν οι Τσέχοι θεωρήσει για να πάνε στον Καναδά. Ε, ε, la parola alla collega Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, πρώτα για την Κροατία και μετά για τη Βοσνία Ζηγοβίνη θα σας ρωτήσω, είπατε πως η Κροατία σημειώνει καλή πρόοδο. Τελεία. Ευτυχώς που ρώτησαν κάποια πράγματα και οι συνάδελφοι Κοιτάξτε, τα εξωτερικά σύνορα δεν είχαν καθοριστεί όταν εντάξαμε τη Σλοβενία. Τώρα που θα γίνουν και εσωτερικά σύνορα αποτελούν εμπόδια για τις διαπραγματεύσεις, πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Νομίζω είναι η πρώτη αποστολή της Προεδρίας να βοηθήσει να λυθεί αυτό το, το πρόβλημα. Άλλο πραγματοκαστήριο, άλλο διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε βεβαίως εσείς ε, και πόσο τεταμένα είναι τα, τα πνεύματα. Για την Βοσνία τα είπαν οι συνάδελφοι, για την Βίζα με την απόφαση που ελήφθη έχουμε ουσιαστικά ε, επιβεβαιώσει τις εθνικές τους εθνικούς διαχωρισμούς και ενισχύουμε τους ακραίους. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε την Βοσνία. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε Βοσνία και Σερβία στο ίδιο τσουβάλι. Πρέπει να βοηθήσουμε να θεραπεύσουμε αυτό το οποίο τελικά έχει καταστραφεί σε αυτή τη χώρα, δηλαδή την συνύπαρξη των εθνοτήτων. Επίσης είπατε πως θα πρέπει να ξεπεράσουν τις παλιές δομές και να οδηγηθούν προς δομές των Βρυξελών. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ κυρία Πακ, ο κύριος Νούνιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι κύριε Μπίλτ, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Τις προάλλες στην παρουσίαση της Σουηδικής Προεδρίας στην Ολομέλεια δεν ακούσαμε πολλά την εξωτερική πολιτική. Το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας και εσείς ε, αναφερθήκατε ρητά τώρα στους προσανατολισμούς που δεν έχουν να κάνουν με την ανατολική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε και περισσότερα, να μας μιλήσετε περισσότερο για τη Λατινική Αμερική και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο θα δώσετε πολιτική όθεση στις διαδικασίες για τις συμφωνίες σύνδεσης με τη Μερκοσούρ και την κοινότητα των Άνδεων. Ξέρω ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει ένας γύρος διαπραγματεύσεων στη Λίμα αυτή την εποχή ε, των άνδρων και θα ήθελα να ξέρω τώρα για την Μεσόγειο φυσικά και θέλω οι ευρωμεσογειακές σχέσεις να ε, βγουν πια από τα προβλήματα και τη σύραξη που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Αυτό ακριβώς θα ήθελα και εγώ. Θα ήθελα τη συμμαχία των πολιτισμών. Μία ερώτηση τώρα για την εξέλιξη των συμφωνιών που έχουμε εδώ προχωράμε καθόλου, έχει αλλάξει τίποτα. Ο συνάδελφος Γκάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε το ότι αυξάνονται οι εντάσεις και Αντί να αντιδρούμε νομίζω καλύτερο θα είναι να δρούμε προληπτικά στις διάφορες περιοχές έντασης και αυτό αφορά και την πολιτική γειτονίας και όσον αφορά την Ουκρανία νομίζω πως είχε λάβει κάποιες αποφάσεις το Συμβούλιο ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα εσωτερικά πρώτα απ' όλα στην Ουκρανία για να μπορέσουμε να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουν να προσεγγίσουν περισσότερο την Ιουνίου. Από ό,τι φαίνεται 18 Ιουνίου οι Υπουργοί Εξωτερικών Σικόρσκι και Στάιν Μάιρο ο συναντήθηκαν στο Κίεβο, ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα. Στόχος είναι... Ποιο στόχο έχετε θέσει όσον αφορά τη σχέση με την Ουκρανία. Μετά είπατε πως θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και στις ε, κρίσεις, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε και καλύτερα προετοιμασμένοι για να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις μας. Πριν από πέντε χρόνια είχαμε αποφασίσει να σχηματιστούν αυτές, αυτές οι μονάδες μάχης ε, ταχείας αντίδρασης οι οποίες δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί σε αποστολές ε, ΚΕΠΑ είχε πάει μια αποστολή της ε, Υποεπιτροπής ε, Άμυνας και Ασφάλειας Σουηδία πέρσι και εντυπωσιάστηκε από την ετοιμότητα της Σουηδικής αυτής ομάδας μάχης. Νομίζω και η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία ήταν προετοιμασμένες αλλά δεν υπήρξε κινητοποίηση στο Κονγκό. Το ερώτημα είναι είστε διατεθειμένοι να ξαναδείτε τις διαδικασίες κινητοποίησης αυτών των μονάδων για να μπορέσουμε τελικά όταν απαιτείται να τις χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. La parola, la collega out. Ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Χάουταλα που είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αμέσως μετά θα απαντήσει ο κύριος Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπίλτ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σε συγχαίρω για το πρόγραμμά σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχω μερικές ερωτήσεις. Θέλετε τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα να είναι πιο εμφανή στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, είπατε. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε πώς θα το πετύχετε αυτό. Πώς θα αυξήσετε το προφίλ αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάλογο με τις τρίτες χώρες, έτσι ώστε να υπάρξουν ορισμένε χρήσιμες συνέπειες παραδείγματος χάρη διαβουλεύσεις με την Κίνα ή με τη Ρωσία. Μετά έχουμε το θέμα της ελευθερίας έκφρασης στο ίντερνετ. Το ίντερνετ, το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου καταστέλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλές αγίδες κατεβάζουν από το ίντερνετ πολλές φορές. Είναι λοιπόν ένα θέμα αυτό. Έπειτα, αυτοί που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, πολλές φορές ε, υφίστανται ε, σοβαρές διώξεις. Στην Ιταλία, Σμυρόβα, παραδείγματος χάρη, δολοφονήθηκε, όπως ξέρετε, με έναν εσχρό τρόπο. Ε, στο φως τη ημέρα, κυριολεκτικά ανοιχτά την δολοφόνησαν. Τι μπορεί να κάνει η Ένωση να βοηθήσει για τα άτομα τα οποία δίνουν μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ενδεχομένως με κυρώσεις κατά χωρών, όπως συμβαίνουν αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και την κυρία Χάτολα. Ο και μετά ο κύριος Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στην πρώτη παρέμβασή σας στην Ένωση για τη Μεσόγειο και αναφερθήκατε σε κάτι που το δεχόμαστε σχεδόν όλοι, ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αναφερθήκατε στη δημογραφική διάσταση, αναφερθήκατε στην οικονομική διάσταση, υπάρχει φυσικά γεωπολιτική, ενεργειακή διάσταση, αλλά η πρωτοβουλία αυτή που πρόσφατα άλλαξε κάπως φαίνεται να έχει βαλτώσει και ερωτώ. Πρώτον, πείτε μας, οι τελευταίες συναντήσεις που έγιναν και δημοσιονομικά και ως προς το περιβάλλον ε, απελευθερώνουν κάπως την κατάσταση, την ελαφρύνουν ώστε να βγει από αυτό τον βάλτο στον οποίο βρίσκεται. Και δεύτερον, στη διάρκεια της Προεδρίας σας σκοπεύετε να πάρετε μια πρωτοβουλία, γιατί θα είναι σημαντικό κάτι τέτοιο, μια πρωτοβουλία για να δοθεί η αναγκαία όθηση στην διαδικασία αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον κύριο Βεγιό. Και τώρα το λόγο πάλι ο κύριος Υπουργός. Σας ευχαριστώ. Ας ξεκινήσω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί όντω είναι προτεραιότητα όχι μόνο της Ουδικής Προεδρίας, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά. Και πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα μέτρα ώστε να ανυψωθεί το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία τους, αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμάμε όλος ιδιαίτερος. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφωνία μεταξύ των Υπουργών αλλά εντάξει, μερικέ φορέ υπάρχουν πράγματα για τα οποία δύσκολα βρίσκουμε ισορροπία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Αποτελεί ηγετική δύναμη. Και περιμένουμε στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά. Που είναι πολλά, σίγουρα. Το διαδίκτυο τώρα. Είναι επίση ένα τρόπο καταπολέμησης των παραβιάσεων υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να περιορίσουν την ελευθερία. Και ίσως δεν ε, τα έχει λάβει υπόψη της η διεθνή κοινότητα που ασχολείται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αρκετά. Εμείς ως Προεδρία φροντίζουμε να ακουστεί η άποψή μας για το Καζακστάν, για παράδειγμα για την νέα νομοθεσία που έχουν εκεί, που περιορίζει πάρα πολύ την ελευθερία στο διαδίκτυο. Στον Πακού ήμουν χτες, με... που κλείσα δύο μπλοκ. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να εξηγήσω. Μερικές φορές είναι άλλος κόσμος, ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν. Ε, τα φροντίζουμε, εν πάση περιπτώσει, όπως μπορούμε. Είναι ένας νέος αγώνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή του μετόπου, οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε μαζί. Και όταν πρόκειται για άλλου είδους προστασίες σε άλλα επίπεδα και σε ατομικό επίπεδο. Έρχομαι τώρα στη Λατινική Αμερική. Δεν αναφέρθηκα σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιπτώσεις, ούτε και στην Αφρική, όπου υπάρχουν πολλά ζητήματα και εκεί, αλλά δεν είχα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου. Η πρώτη διάσκεψη που θα έχω είναι με την Βραζιλία και η Βραζιλία είναι ένα σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Όχι μόνο όσον αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ, την ενέργεια, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα. Οι Ονδούρε επίση είναι ένα από τα θέματα τα οποία ε, συζητάμε με τη Λατινική Αμερική επί του παρόντος. Σίγουρα όταν πρόκειται για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου είμαστε πολύ δραστήριοι και προσπαθούμε να ελέγξουμε την κάθε λεπτομέρεια. Με την κοινότητα των Άνδεων είμαστε σε επαφή. Έχουμε το θέμα της Κεντρικής Αμερικής που είναι λιγάκι σε εκκρεμότητα, αλλά ελπίζουμε να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε και αυτό. Έτσι ενισχύονται οι σχέσεις μας με τις αναδυόμενες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής. Αυτά τα θέματα για να ξανάρθουμε σε προηγούμενα ζητήματα. Κοιτάξτε, επειδή μιλήσαμε για τη Βοσνία πριν, αυτά τα ζητήματα δεν τίθεται μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Σας ξαναλέω ότι ήμουν στον Πακού χτες. Άλλη χώρα. Εντάξει. Αλλά πάλι είναι θέμα ε, συμφωνίας εταιρικών σχέσεων. Περισσότερες πτήσεις υπάρχουν ανάμεσα στη Μόσχα και τον Πακού σήμερα από ό,τι υπήρχαν την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει θεώρηση. όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άνθρωποι από τη Γεωργία, τη Συρία λοιπά θέλουν ελευθέρωση των θεωρήσεων. Ελπίζουν, ονειρεύονται. Οι Ουκρανοί το θέλουν. Για να δούμε. Δεν είναι αυτονόητο. Αυτά είναι δύσκολα ζητήματα. Εγώ πολύ θα ήθελα να ανοίξουμε όσο γίνεται περισσότερο και πιστεύω στην καλή θέληση όταν οι άνθρωποι συμβρίσκονται, γνωρίζουν οι μεν τους δε, λύνονται πολλά προβλήματα, αλλά υπάρχουν και εσωτερικά ζητήματα. Ορισμένοι έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς, Δεν μιλάω εδώ για τους υπουργού εσωτερικών, αλλά υπάρχουν και τα θέματα εγκληματικότητα, ηλεθρεμπορίου ή άλλα. Οπότε εκεί μπαίνει πρόβλημα και δημιουργείται και πολιτικό ζήτημα μεταξύ των χωρών μας. Σας είπα, είναι δύσκολο να βρούμε την ισορροπία. Θέλουμε να ανοίξουμε τα σύνορά μας όσο γίνεται πιο γρήγορα για όσο γίνεται περισσότερες χώρες, αλλά συγχρόνως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το θέμα της καταπολέμησης, της εγκληματικότητας, του λαθρεμπορίου, της εμπορίας παιδιών, γυναικών, οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει συγχρόνως να είμαστε και προσεκτικοί και αυστηροί να ελέγχουμε την ταυτότητα του καθενό. Αλλά θέλω να προχωρήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα και να ανοίξουμε ε, τις χώρε μα όσο γίνεται περισσότερο. Σίγουρα τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν την προτεραιότητα, αλλά βλέπετε είναι πιο εύκολο για τη Ρωσία από ότι για τη Γεωργία. Ή για τη Ρωσία από ότι για την Ουκρανία. Είναι σωστό. Ε, δεν μπορεί να το πει αυτό κανείς. Πώς να αλλάξει. Είναι μία ερώτηση με την οποία πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές τους Βόσνιους. Τους βοηθάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να τους βοηθάμε. Αλλά πρέπει και εκείνοι να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Τι θέλω να πω ε, με αυτό. Ωραία, όλοι στρέφονται προς τις ε, Βρυξέλλες. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό. αλλά πρέπει να δούμε πώς θα ερμηνευτεί και η συμφωνία. Ξέρω την έχω διαπραγματευτεί και εγώ, αλλά το Dayton δεν φτάνει έτσι κι αλλιώς για τη Βοσνία. Είναι η αρχή. Τώρα πρέπει οι Βόσνοι να δράσουν. Και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Αν συγκρίνουμε τι λέει η Νευτική Συμφωνία Dayton και μετά, με το κοινοτικό κεκτημένο, δεν τίθεται θέμα, το κοινοτικό κεκτημένο είναι αυτό που βοηθάει και την κοινωνία της Βοσνίας να αλλάξει και να εξυγχρονιστεί όλο και περισσότερο. Γι' αυτό και η μετάβαση πρέπει να γίνει όταν γίνεται από τις δομές της προσανατολισμένες των τέτων προς τις δομές εκείνες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν πλήρη μέλη και να μπορούν να ανταποκριθούν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι πιο απαιτητικό, αλλά και θα βοηθήσει τη Βοσνία να σταθεροποιηθεί περισσότερο. Τα συζητάμε αυτά με τις αρχές της Βοσνίας. Με τους φίλους, με τους εταίρους μας, Τουρκία, Ρωσία για παράδειγμα. Τέλος, για την Ισλανδία και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ναι, τα ξέρω λίγο εδώ τα πράγματα, γιατί θυμάμαι ότι και εμείς όταν ε, ζητήσαμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περάσαμε από αυτό. Πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευτούμε ε, την ε, ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρώτα ήταν το θέμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ένα πρόβλημα ήταν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε τότε το Μάστριχτ που δημιουργούσε ταραχές. Λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η βάση για την ένταξη στη συνέχεια. Η Ισλανδία το έχει προχωρήσει αυτό και η Νορβηγία και το Λιχνιστάιν. Για να πάρουμε για παράδειγμα αυτές τις τρεις χώρες. Που σημαίνει ότι όποια από αυτές τις τρει χώρες ζητήσει να ενταχθεί, έχει ήδη καλύψει ένα μεγάλο μέρος του δρόμου. Φυσικά μένουν και άλλα σημαντικά ζητήματα, δεν λέω, αλλά ο κύριος όγκος των διαπραγματεύσεων θα έχουν ήδη καλυφθεί, σας το λέω, από εμπειρία που έχω από τη Σουηδία, από την Αυστρία, τη Φιλανδία, γιατί και εμείς πήγαμε τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νορβηγία δεν προχώρησε, η Ισλανδία δεν ζήτησε ποτέ Αν υπάρχει προοπτική αυτό για άλλους, ε, τι να σας πω, θέλω να είμαι θέλω να πιστεύω σε αυτή τη δυνατότητα, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Διαπραγματευόμαστε κυρίως με την Ουκρανία για το ελεύθερο εμπόριο. Τώρα αν έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί και αυτοί στην Ουκρανία στα εσωτερικά τους έχουν πολλά ζητήματα. Ε, πάντα, ή τέλο πάντων συχνά η δημοκρατία έτσι είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρώτα πρέπει να δούμε με τη συμφωνία αυτή. είναι στο ελεύθερο εμπόριο προ τα τέλη τη χρονιά. Είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι είναι εφικτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά, ίσω, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και με τη Γεωργία. Και ίσω και με άλλου. Και έτσι ίσως δημιουργηθεί μια περιοχή, ένας χώρος που να οδηγεί σε μια εσωτερική αγορά. Ίσως. Θα δούμε. Το αν θέλουμε να τους εμποδίσουμε, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά λέω ότι αν αυτό γίνει, θα διευκολυνθεί η διαδικασία. Τα πράγματα πρέπει να πάνε με τη σειρά. Μην προτρέχουμε. Οπότε εγώ χαίρομαι για τα μικρά βήματα που κάνουμε όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο και μετά θα δούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κάνω έκκληση στην κατανόησή σας. Έχουμε 30 λεπτά και 20 παρεμβάσεις. Μοιραία ο κάθε ομιγητής θα πρέπει να μην ξεπεράσει το ένα λεπτό. Πρώτος ο κύριος Κουκ... Α, μια ερώτηση. Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ σήμερα. Με ευχαρίστηση διαπίστωσα ότι η διεύρυνση η συνεχόμενη, συνεχιζόμενη διεύρυνση συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητές σας. Νομίζω ότι η προσωπική σας εμπειρία θα πρέπει να χρησιμεύσει σαν ένα μπόνους. Με όλη την εμπειρία που έχετε κύριε Υπουργέ, στα Βαλκάνια, επί έτη, μην είστε μετριόφρονο, δεν χρειάζεται να είστε μετριόφρονο μεταξύ μας. Θεωρώ ότι η Σουηδική Προεδρία στο πρόσωπό σας και η τρέχουσα κατάσταση στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι δύο πράγματα πάρα πολύ συμβατά μεταξύ τους και όρος Ευρωπαϊκή Προοπτική που είναι το πιο ισχυρό κίνητρο για τις χώρες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσά. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό παρακαλώ. Πρώτα σας ευχαριστούμε κύριε Κούκαν. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος Μποντί. Κύριε Υπουργέ, χθες το βράδυ στην τηλεόραση, ίσως να το είδατε, βλέπαμε εικόνες από μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Τουρκία. Η Τουρκία γιόρταζε την επέτειο της εισβολής στην Κύπρο και της κατοχής της Κύπρου μια κρίση που συνεχίζεται όχι εδώ και 20 χρόνια, εδώ 35 χρόνια. 35 χρόνια που ένα κομμάτι, σχεδόν το μισό, της ε, χώρας αυτής που είναι μέλος της Ένωσης βρίσκεται υπό κατοχή. Ποια είναι η εκτίμηση σας κύριε Υπουργέ για τη γιορτή αυτή στην Άγκυρα. Δεν έρχεται σε αντίφαση με την υποψηφιότητα που έχει υποβάλει. Με άλλα λόγια, μια χώρα μπορεί να είναι υποψήφια για ένταξη στην Ένωση ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας δόξα για τον εαυτό της το ότι εισέβαλε και κατέχει στρατιωτικά ένα τμήμα μιας χώρας μέλους της Ένωσης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε Μποντή. Τώρα ο επόμενος άλλος αντιπρόεδρος, ο κύριος Πασκού. Αν θεωρήσουμε επιτυχία στο Αφγανιστάν σε σχέση με αυτό που αφήνουμε πίσω μας όταν φεύγουμε και αν ξεκινήσουμε από το ότι η άμαχη, ο άμαχος πληθυσμός είναι η, η μη στρατιωτική μάλλον συνιστός είναι πιο σημαντική από τη στρατιωτική είναι λογικό να περιμένουμε μια πρωτοβουλία για να έχουμε περισσότερη ακολουθία και συνοχή και δυναμισμό στην προσπάθεια της Ένωσης προκειμένου να υπάρξει ένα σωστό θεσμικό καθεστώς εκεί. Πρώτα, σας ευχαριστούμε τον κύριο Πασκού, ο κύριος Βάλτερ. Η κυρία Βάλτερ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω για την ε, στρατηγική σένα της Ρωσίας, για τη Βαλτική, και για την γεωργία. Πώς θα πετύχετε τη συμφωνία των έξι σημείων. Αυτό θα ήθελα να πω, αλλά θα κάνω μια ερώτηση που αφορά το άμεσο μέλλον. Όπως ξέρετε, πρέπει ένα χρόνο το Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε όλα τα εθνικά κοινοβούλια να αναγνωρίζουν την 23η Αυγούστου ως κοινή μέρα ανάμνησης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού. Ξέρω ότι λίγα εθνικά κοινοβούλια ήδη εισήγαγαν αυτή την ημέρα με αυτά τα χαρακτηριστικά και θέλω να ρωτήσω η Σουηδία τι έκανε. Και σκοπεύετε να ενθαρρύνετε τους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο να το κάνουν, να αναγνωρίσουν δηλαδή την κοινή αυτή ημέρα γιατί πλησιάζει αυτή η θλιβερή επέτειος του, της συμφωνίας του συμφώνου Χίτλερ-Στάλιν. Ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη νότια όχθη της Μεσογείου. Αυτό που γίνεται στην Κύπρο και για την Τουρκία το ανάφερε οι συνάδελφοι. Η Αλγερία είναι μια χώρα όπου δόθηκαν μάχες όπως και στο Ιράκ με πάρα πολλούς νεκρούς παρόμοια με το νούμερο που έχουμε στο Ιράκ. Στη Λιβύη, στο Λίβανο, έχουμε φαινόμενα που έχουν επιπτώσεις με τον τρόπο τους στη ζωή του ευρωμεσογειακού σεναρίου και ρωτώ. Υπάρχει στρατηγική της Ένωσης για το ευρωμεσογειακό σενάριο. Τα προβλήματα που όλες αυτές τις χώρες δεν θα μπορούσαν να γίνουν πιο καλά κατανοητά και να επιληθούν αν τα αξιολογήσουμε μέσα στα πλαίσια ενός περιφερειακού σενάριου. Και αυτό το περιφερειακό σενάριο είναι η πραγματική πρόκληση για το μέλλον για την Ευρώπη. Υπήρξαν συγκεκριμένες δράσεις όσον αφορά το σενάριο για την Ανατολή, αλλά φαίνεται να μην υπάρχει ένα όραμα σχετικά με το τι θέλουμε να πετύχουμε ως προς τον Νότο, Πρόεδρος ο κύριος Κάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, υποστηρίζω τις προτεραιότητες που αναφέρατε. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα ο παγκόσμιος ρόλος της Ένωσης. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας για να βελτιωθεί η δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων. Δεύτερον, τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομίζω φυσιολογικό είναι να βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Το ζήτημα αυτό εννοώ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμέσως ενθαρρύνει διαχωρισμό με βάση τις εθνοτικές γραμμές στην Βοσνία, κάτι το οποίο θέλουμε όλοι να αποτρέψουμε. Και δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον σερβικό και τον κροατικό πληθυσμό της Βοσνίας να πάνε στο Βελιγράδι και στο Ζάγκρεμπ για να πάρουν διαβατήρια για να μπορούν να μπουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βρούμε νέους τρόπους για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση του Σεράγεβου να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Η πρότασή μου λοιπόν για σας κύριε Πρόεδρε και Λεμπερτίν είναι η εξή. Ας προσκαλέσουμε τον ειδικό απασταλμένο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τον πρέσβη τον κύριο Ίνσκο, το στομότερο δυνατόν για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων εδώ για την κατάσταση και τα καλύτερα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τάλε. Ευχαριστώ κύριε Τάλε. Παρακαλώ του ε, συναδέλφους που θα μιλήσουν να σέβονται το χρόνο. Κυρία Γιαννάκου. Ε, κύριε Πρόεδρε, στην, ε, στο πρόγραμμα της Προεδρίας, το οποίο πραγματικά βρίσκω ότι είναι εξαιρετικό, ε, μιλάτε για την ασφάλεια και την άμυνα και τη συνδέεται με την ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Δίνεται δε ιδιαίτερη έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τη δημοκρατία. Λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανσή σας σχετικά με τον πρόεδρο Ομπάμα, πώς νομίζετε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να αναδιοργανωθεί ο τομέας ασφάλεια και άμυνα προς την κατεύθυνση μιας πιο συγκροτημένης διεθνούς παρουσίας της Ένωσης στην υπόθεση της διαχείρισης κρίσεων ιδιαίτερα δε στο τμήμα συνεργασία για ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννάκο. Περνάμε στους φιλελεύθερους. Βάγκελ. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω πως είστε πολύ ενεργός και και θα εκμεταλλευτείτε σίγουρα το χρόνο που έχετε ως προεδρεύον του Συμβουλίου. Φαντάζομαι είναι φρικτό να, να ζει κανεί στα ερήπια της Γάζας αυτή, αυτή τη στιγμή και στις αφύσικες συνθήκες αυτού που θεωρείται Παλαιστινιακό κράτος. Πρέπει να αναμειχθούμε ενεργά, να προσπαθήσουμε να επανεκκινήσουμε αυτή τη διαδικασία και να έχουμε αξιόπιστη ευρωπαϊκή πολιτική στη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, θα ήθελα να σας επενέσω για την μετριοπαθή σας στάση στην διαμάχη Σλοβενίας-Κροατίας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε στα βήματα του Όλη Ρεν. Ήταν καλή η πορεία που έχει χαράξει. Χρειάζεται συμβιβασμός και, στις δύο, και από τις δύο πλευρές. Σπάνιο πράγμα βέβαια η διάθεση για συμβιβασμό, αλλά ελπίζω να τα καταφέρετε. Ευχαριστώ. Bene, eh, ευχαριστούμε. Πριν τον Υπουργό, η συνάδελφος Φλότρα, πρώην πρόεδρο τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. σα παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλή σα μέρα κύριε Μπίλτ. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τη Λιβύα. Ακούμε, εδώ είμαι, εδώ είμαι, με βλέπετε. Μιλάμε λοιπόν ε, για την υπογραφή μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Λιβύα στα τέλη της χρονιάς, δηλαδή υποσυνδική προεδρία. Προεδρίας. Σε τι πλαίσια γίνεται η διαπραγμάτευση τη συμφωνία αυτή, μια που δεν αποτελεί μέρο ε, τη διαδικασία τη Βαρκελόνη η Λιβύα, και πώ θα συμπεριλάβετε τα ανθρώπινα δικαιώματα στι ε, διαπραγματεύσει για τη συμφωνία αυτή με τη Λιβύα, μια που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ξέρουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στη Λιβύη. Έπειτα γιατί η Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση λέτε ότι θα στηρίξετε και ελπίζετε ότι είσαστε αισιόδοξο όσον αφορά την Προεδρία σα για το ε, κατά πόσο, κατά διάρκεια τη Προεδρία σα θα επιτευχθεί συμφωνία στην Κύπρο και λέτε ότι θα τη στηρίξετε, αλλά αυτό έχει να κάνει και με άλλη υποχρέωση του Συμβουλίου που είναι να φροντίσει για την πρόσβαση στου λιμένες. Εδώ υπό την Προεδρία σα θα μπορούσατε να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Εσείς αυτή την προοπτική πώς τη βλέπετε. Ευχαριστούμε. Ο υπουργό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Πράγματι είπα πως ως Προεδρία θα ακολουθήσουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Είναι πολλές που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα. Δεν σχετίζονται συνδέονται μεταξύ τους, πρέπει να τις δούμε όμως σε ένα πλαίσιο. Σας διαβεβαιώ λοιπόν πως εξτάζουμε προσεκτικά όλα τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει για την εφαρμογή. Την εφαρμογή τους πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την Κύπρο. Για την Κύπρο λοιπόν. Ε, μιλήσατε για πράγματι την εισβολή ενός κράτους μέλους το 1974. Ο κύριος Παπαδόπουλος νομίζω δεν ήταν πια επικεφαλής της Χούντας. Κάποια απεχθής φιγούρα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πολύ διπλωματική η δήλωσή μου. Η Χούντα λοιπόν στην Αθήνα ήταν αυτή που ξεκίνησε τα γεγονότα που οδήγησαν τελικά σε αυτά Βεβαίω δεν επρόκειτο τότε για κράτο μέλο, δεν, δεν μπορούσε να πλησιάσει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχοντα. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν έχει γίνει τίποτα έκτοτε και πράγματα τα οποία θα ήταν δυνατά το 2004 όταν γίνονταν κράτος μέλος η Κύπρος δεν έγιναν και ξέρουμε γιατί δεν έγιναν και είναι η κληρονομιά της δεκαετίας του 60, του 74, του 2004 ε, που έχουμε τώρα. Και πάρτε όποιο κομμάτι αυτής της κληρονομία θέλετε εσεί, αλλά ε, έχουμε όλη αυτή την κληρονομιά τώρα να αντιμετωπίσουμε. Οπότε ε, δεν ανάγκη τώρα να δίνουμε τις μάχες του παρελθόντος, πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Έχουμε δύο ηγέτε στην Κύπρο, τον πρόεδρο Πιστόφια και τον κύριο Ταλάτ, που είναι πεπισμένοι και σκοπεύουν να ξεπεράσουν όλα τα προβλήματα του παρελθόντος. Ε, ας ελπίσουμε ότι θα επιτύχουν. Και με κάθε τρόπο που μπορούμε θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε και ως άτομα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την Νήσο, είναι για την περιοχή ολόκληρη, αλλά και για να δείξουμε πως ε, υπάρχει προσήλωση στα ευρωπαϊκά ιδεώδη, δηλαδή να ξεπερνάμε τις συγκρούσεις και τους πολέμους του παρελθόντος και πράγματι, όπως όλοι ξέρετε, είχαμε πολλούς τέτοιους στο, στο παρελθόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και στο συγκεκριμένο τμήμα. Για τη Μέση Ανατολή συμφωνώ πλήρως πως πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή, κάτι βεβαίως το οποίο εύκολα λέγεται αλλά δύσκολα γίνεται. Το καλό είναι ότι Τώρα είτε δεν ξέρω αν εμείς μιλάμε αμερικάνικα ή ή ευρωπαϊκά, αλλά μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ε, εδώ και καιρό. Και έχουμε και ουσιαστικό διάλογο με τη νέα Ισραηλινική κυβέρνηση σε πολλά σημαντικά ζητήματα. Αποδίδουμε σημασία στην νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία. Υπάρχει μια πρωτοβουλία, υπάρχει κατάσταση που είναι προβληματική στις ε, παλαιστινιακές περιοχές και από οικονομική και από πολιτική πλευρά και Πρέπει να ξέρετε πως ε, τον Ιανουάριο του επομένου έτους, ε, ίσως και λίγο αργότερα, θα έχουμε εκλογές στην Παλαιστίνη και είναι σημαντικό το ποιος θα κερδίσει αυτές τις εκλογές. Θα κατέβουν στις εκλογές όλες οι δυνάμεις ε, των Παλαιστινιακών περιοχών και αυτές που μας αρέσουν και αυτές που δεν μας αρέσουν. Έτσι είναι οι εκλογές και ελπίζω να δημιουργηθεί κάποια ελπίδα για την ειρηνευτική διαδικασία στους μήνες πριν τις εκλογές ε, για να επηρεαστεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε και εμείς στην ευρωπαϊκή πλευρά. Γνωρίζω πως το έχουν υπόψη τους και στην Ουάσιγκτον. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Ε, υπάρχει και ο Λίβανος, θετικές εξελίξεις εκεί. Είμαστε σε διάλογο με τη Σύρια. Είναι πολλά ζητήματα επιτάπητος ε, για ολόκληρη την περιοχή και το, το Παλαιστινιακό βεβαίω είναι κρίσιμο. Κάποια ερωτήματα δεν τα απάντησα πριν. Ένα ήταν για την Τσεχία και την Βίζα. Εμείς ε, ζητήσαμε από την Κομισιό να μας πει τι, γίνεται γιατί είναι ζήτημα της Κομισιόν. Θα δούμε τι θα, πώς θα αντιδράσουμε. Κατόπιν έχουμε τα διαφορετικά ζητήματα της ομάδες μάχης, τις ε, δυνατότητες ε, αντιμετώπισης κρίσης, το ανέφερε και η κυρία Μαργίδα Γιαννάκου. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος ε, διαχείρισης κρίσεων και δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχουμε δει τώρα τι γίνεται με την εκείνη μας Προεδρία, με τους Τσέχους και, τους, ε, και τη δική μας τώρα τη Σουηδική. Υπάρχει πράγματι πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, ανάγκη, αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο μία από τις εξαμήνες ε, προεδρίες ε, με... Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Έχουμε επιστήματα τη επιτυχία μας. Οπότε πρέπει να έχουμε καλύτερα θεσμικά όργανα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση που υπάρχει για ευρωπαϊκή παρέμβαση ανά τον κόσμο και πράγματι να έχουμε και καλύτερες δυνατότητες και διπλωματικές και βοήθειας και αμυντικές. Ένα κομμάτι αυτών είναι οι μονάδες μάχης. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να δω, καλά βεβαίω αυτό είναι ζήτημα υπουργών μείνεις όχι εξωτερικών, θα ήθελα να δω αν υπάρχουν πράγματι. Ε, Τέλο δεν είναι πολύ διπλωματικό αυτό που λέω γιατί σε μια άλλη επίσκεψη από αυτήν που αναφέρατε ε, είχαμε λόγους να αναρωτηθούμε αν υπάρχουν όντως αυτές οι ομάδες μάχης. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν σε κάποιο χαρτί στις Βρυξέλλες, αλλά το τι γίνεται επί τόπου, αυτές οι μονάδες ήταν ή αλλού ή πουθενά. Και πρέπει να το δούμε αυτό. Πράγματι πρόκειται για ένα μέσο που έχουμε ένα ακριβό μέσο, το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούνται δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παραπονόμαστε πολύ. Η Σουηδία έχει ένοπλες δυνάμεις, έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και δεν τις έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ και 150 χρόνια. Αυτό είναι καλό. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα τις καταργήσουμε. Ε, οπότε το ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις ομάδες μάχης δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις έχουμε. Απλά πρέπει να υπάρχουν, ώστε όταν χρειαστούν, ελπίζουμε όχι, αλλά όταν χρειαστούν θα είναι διαθέσιμες και θα μπορούν να αναπτυχθούν σε 10 μέρες. Μαζί με τις, ε, τους πόρους που θα έχουμε από πλευράς ε, διπλωματίας, ε, βοήθειας κλπ. Και πρέπει πράγματι να υπάρχει ετοιμότητα στις Βρυξέλλες. Τώρα για την Μεσόγειο και τη συνολική στρατηγική. Αυτό υποτίθεται πως είναι η Ένωση της ε, Μεσογείου. Με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, εγώ είμαι υπέρ της έννοιας ε, αυτή. Γνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτές είναι οι δυσκολίες της Ένωσης, αλλά υπάρχει και ένα φιλοσοφικό ζήτημα. Και το ίδιο ισχύει επί τη ευκαιρία και για την ανατολική εταιρική σχέση. Είναι μία εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης συνολικά και της συγκεκριμένης περιοχής. Οι Βρυξέλλες, δηλαδή και 27 ε, που ασχολούνται με τα ζητήματα της Μεσογείου. Εξού και η προσθέμενη αξία της Ένωσης δεν είναι μόνο οι χώρες της Μεσογείου που καλώ κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά η Ένωση συνολικά. Το ίδιο και με την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Δεν είναι ζήτημα Σουηδία και Πολωνίας. Είναι εταιρική σχέση ολόκληρης τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των θεσμικών οργάνων τη με τι χώρε αυτές. Και όταν το λέω έτσι βεβαίως αυτό έχει κάποιες ε, συνέπειες για τη θεσμική μας λειτουργία. Αλλά μακροπρό νομίζω έτσι θα διαμορφωθούν και θα μεταμορφωθούν αυτές οι σχέσεις και οι χώρες ε, και αυτό είναι που αναζητούμε. Για την 23η Αυγούστου και το Σουηδικό Κοινοβούλιο η απάντηση είναι δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά είναι κάτι που θα γίνει νομίζω Ειλικρινά δεν ξέρω. Το πρόβλημα είναι βεβαίως πως το Σουηδικό Κοινοβούλιο ε, βρίσκεται σε βαθιές διακοπές εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως τίποτα δεν αποκλείει το να συμβεί κάτι. Αλλά υπάρχουν διαφορετικές ε, ημερομηνίες ε, που ακολουθούν τους ερχόμενους μήνες μίλησα για το να, να κοιτάμε προς το μέλλον. Βεβαίως καλό είναι να θυμόμαστε και το παρελθόν. Υπάρχει πράγματι, όπως είπα, η 10η Αυγούστου, η 23η, η 1η Σεπτεμβρίου, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, η 9η Νοεμβρίου και η 17η Νοεμβρίου. Για να σκεφτούμε το τι συνέβη στο παρελθόν και το τι συνέπειες έχει αυτό για το μέλλον. Και την οικοδόμηση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν τώρα και τι προτεραιότητε. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να επανέλθουν, εννοώ την Γραμματεία του Συμβουλίου και την Κομισιόν να έρθουν και να ενημερώσουν του Υπουργού Εξωτερικών τον Σεπτέμβριο για ένα ενισχυμένο πακέτο για το τι μπορούμε να κάνουμε από πλευρά ε, πολιτική μη στρατιωτική και διπλωματική στο Αφγανιστάν για να συμπληρώσουμε τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε και την ειρήνη, αν θέλετε, για να υπάρχει σταθερότητα στο Αφγανιστάν στο μέλλον και μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερους από τους ε, πιο διευρυμένους πόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον, αλλά όλοι ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την κινητοποίηση. Αλλά υπάρχει οπωσδήποτε φιλοδοξία. Και τέλος αναφέρατε κύριε Κουκ την ευρωπαϊκή προοπτική. Πράγματι είναι κάτι που με εντυπωσιάζει πάντα το τι δύναμη έχει. Αυτό μπορεί να ισχύσει στα Δυτικά Βαλκάνια, στο Νότιο Κάφκασο, στην Ουκρανία. Εμείς, εσείς ως βουλευτές εκπροσωπείτε ένα όνειρο για πάρα πολλές χώρες εκτός των συνόρων μας. Ε, αυτό το όνειρο έχει μία δύναμη να μετασχηματίζει κοινωνίες και αν δεν ε, υπάρχει αυτό το όνειρο, φοβάμαι πως θα κυριαρχήσουν άλλες δυνάμεις και ίσως εφιάλτες. Οπότε για την περιοχή γύρω από την Ένωσή μας είναι πολύ σημαντικό για αυτούς και για τη σταθερότητά μας και οπωσδήποτε η Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια περιοχή κλειδί. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε κύριε Παργιά. Έχουμε ακόμα 10 συναδέλφους που ήθελαν να μιλήσουν. Ο κύριος υπουργό ήδη έχει ξεπεράσει το χρονικό όριο που είχε. 30 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ, Έχει σχόλια, μόνο ερωτήσεις. Προτασχέβιτς. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν σας εκτιμώ ιδιαίτερα για την, το ρόλο σας στην εταιρική σχέση με την Ανατολία. Αλλά έχουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία που καλύπτεται από την ε, εταιρική αυτή σχέση και συμφωνία. Όπως και όπως ξέρετε, 11 ε, άτομα σε ειρηνική διαδήλωση κρατούνται ακόμα στη φυλακή και ο τελευταίος μάλιστα έφαγε ένα χρόνο φυλακή. Τρεις άλλε, τρία άλλα στελέχη ε, κρατούνται και εν αναμονή δίκης σας παρακαλώ βάλτε προτεραιότητα στην πολιτική σας ατζέντα στις σχέσεις με τη Λευκορωσία το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ε, φυλάκισης ε, συγκεκριμένων ατόμων. Η συνάδελφος Κέιζερ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπίλτ, ίσως να μην μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα στη μέση Ανατολή, ωστόσο ε, έχουμε τη Συρία, την αναφέρετε και εσείς, είναι σημαντικό για τη σχέση μας με το Λίβανο, με το Ιράν και με την Παλαιστίνη ενδεχομένω. Η συμφωνία σύνδεση έχει παγώσει. Ο Σαρκοζή κάπως την ξανακίνησε, η Τσεχική Προεδρία κάπως την πάγωσε, σκοπεύετε να το ξανακινήσετε το θέμα αυτό. Ε, είναι στην ημερήσια διάταξη της 4 ε, η και 5 Σεπτεμβρίου. Πρόεδρος. Ο κύριο Κουμουτσάκος. 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Ε, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν κατενόησα στην προηγούμενη απάντησή σας αν η ιστορική σας αναφορά στην ελληνική δικτατορία ήταν μια απόπειρα δικαιολόγηση της 35 χρονη κατοχής, παράνομης κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή δεν ήταν πολύ σαφέ, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό και χρήσιμο να το εξηγήσετε ή, εν πάση περιπτώσει, να το αποσαφηνίσετε στην επόμενη παρέμβασή σας, τώρα που ξεκινάει η Προεδρία της, Σουηδικής, της Σουηδίας. Όσο λάθος είναι, κύριε Υπουργέ, να εκπέμπουμε αρνητικά μηνύματα προς την Τουρκία όταν λέγεται ότι δεν έχει προοπτική να γίνει πλήρε μέλο τη Ένωση, εξίσου λάθο μηνύματα είναι να είμαστε πολλέ φορέ περισσότερο από όσο πρέπει επίοικοι μαζί τη όταν δεν τηρεί τι δεσμεύσει και τι υποχρεώσει τη. Ευχαριστούμε. Παντσέρι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση. Επειδή με ανησυχεί ιδιαίτερα το θέμα της συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την απόφαση του Γερμανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου περισσότερο από το δημοψήφισμα για την Ιρλανδία, σας ερωτώ, αν δεν έχουμε τη συνθήκη σε σχέση με τη διεύρυνση της Ευρώπης. Το σκέφτεστε καθόλου το θέμα. Η απουσία συνθήκης δεν θα έπρεπε να θέσει το πρόβλημα της διεύρυνσης ως κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να υπάρξει μια περίοδος περισυλλογής σε σχέση με την διεύρυνση και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Βαν Μπάλεν, φιλελεύθερη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν για την Κύπρο και από Κύπριος, αλλά θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έχουμε τη Συμφωνία της Άγκυρας και βάσει τη συνθήκη της Βιέννης για τις συνθήκες αυτό σημαίνει ότι τον υπογράψει μια συμφωνία πρέπει να την επικυρώσει και να την υλοποιεί. Πώς στη Φιλοσοφική Προεδρία θα φροντίσετε η Συμφωνία τη Άγκυρας να ε, εφαρμόζεται και από την Τουρκία. Μπότσκουρτ. Ευχαριστώ. Δύο σύντομε ερωτήσει προ τον Υπουργό. Πρώτα απ' όλα για την Τουρκία. Στα πλαίσια της ε, χρονιάς που ξεκίνησε μετά το ατύχημα στο αεροδρόμιο έγιναν διάφορα, ακούσαμε για την Κύπρο επίσης. Λοιπόν, είπατε ότι εξαρτάται από αυτούς. Αν είναι έτοιμοι, περιμένουν, θα δούμε, εξαρτάται πότε θα είναι έτοιμοι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι για τις Ονδούρες. Υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στις ε, Ονδούρες και έχουν αποτύχει το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα πάτε εσείς ώστε να προσπαθήσετε να βρείτε μια λύση εκεί. Λοχ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Μπίλτ. Υπογραμμίσατε πως θέλετε να ενισχύσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τα φέρετε στο προσκήνιο, είναι αναγκαίο, σας υποστηρίζουμε, γιατί η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει υποστεί πλήγμα, καθώς ε, και κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα στην καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Βλέπουμε πως η Αμερικανική κυβέρνηση τώρα διδάσκεται από τα λάθη της και δίνει εγγύηση πως δεν θα συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Το ερώτημά μου είναι σε εσάς τι σκοπεύει να κάνει η Σουηδική Προεδρία έτσι ώστε και τα ευρωπαϊκά κράτη να αναλάβουν την ευθύνη τους για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της της τρομοκρατίας που έχουν ήδη καταγραφεί επαρκώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για το ότι ήρθατε σήμερα εδώ. Η ερώτηση, η ερώτηση μου αφορά την, ε, την θέρμανση της γης και τη συνάντηση των G13. Δεν υπήρξε συμφωνία για τη διαδικασία μετρίασης όσον αφορά τη θερμοκρασία η πρότασή μας είναι, είναι πολύ ευρωκεντρική και δεν υπάρχει μια ε, συγκεκριμένη ρήτρα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό, διότι αν δεν το έχουμε αυτό δεν θα υπάρξει συνολική συμφωνία και τη χρειαζόμαστε απεγνωσμένα τη συνολική αυτή συμφωνία. Ο κύριος Μαυρονικόλας. Συγχαρητήρια για την Προεδρία, για την ανάληψη της Προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουμε στο Κυπριακό δεν μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στις συνομιλίες. Από την άλλη όμω ελέγχει την πορεία ανένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε η Προεδρία να συμβάλλει στο να υποδείξει στην Τουρκία ότι η λύση πρέπει να είναι εντός ευρωπαϊκού κεκτημένου Δεύτερον, ότι η Τουρκία πρέπει να μειώσει την κατοχική της παρουσία στο νησί και τρίτο, αφού μιλούμε για το πρόβλημα της μετανάστευσης και της λάθρομετανάστευσης, θα μπορούσε η Προεδρία να υποδείξει την ανάγκη να σταματήσει ο επικισμός της Κύπρου από την Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. La parola all'onorevole Howitt. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια κύριε Πίλτ για αυτά που μας είπατε και για τις προσπάθειες που έχετε κάνει για τους Βρετανούς στο Ιράν. Για την Γεωργία, δεν ξέρω εσείς συμφωνείτε με την εντύπωσή μου ότι από όσο ξέρω στα πλαίσια των σχέσεων με την Ρωσία, όχι Σοβιετική Ένωση βέβαια, Ρωσία, προβλέπετε να προχωρήσει καθόλου η αποστολή σας όσον αφορά την Αφχασία και τον Κάφκασο. Τελευταία παρέμβαση για τη σημερινή συζήτηση η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Ακούμε μόνο τον Πάπα να μιλάει για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου. Εσείς η δικιά σας η Προεδρία θα κάνει τίποτα στο επόμενο για το Συμβούλιο ασφαλεία του ΟΗΕ. Εσείς θα κάνετε τίποτα γι' αυτό. Έπειτα για τα θέματα ασφάλειας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι το πιο βασικό στο Ιράν. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό. Είσαστε υπέρ. Συγγνώμη από του που θα ήθελαν και αυτοί να μιλήσουν, αλλά χρησιμοποιήσα ένα αυστηρό κριτήριο. αυτός που ζήτησε το, λόγο στην αρχή το πήρε. Για τους υπόλοιπους που καθυστέρησαν, δυστυχώ ο χρόνο δεν υπήρχε, ο υπουργό δεν μπορεί να καθίσει άλλο. Του δίνω το λόγο για το να κλείσει με απαντήσεις στις τελευταίες ερωτήσεις. Τώρα θα είμαι όντω πάρα πολύ σύντομο. Η Ευρωπαϊκή Φωνή για τη Μεταρρύθμιση του Συμφωνίου Ασφαλεία. Απούσα. Διότι υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ απόψει. Υπάρχει διαίρεση στην Ένωση. Μερικοί είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία, έχουν μια αλφα άποψη. Άλλοι έχουν άλλη άποψη. Υπάρχει διαίρεση στι απόψει όσον αφορά τη Συμβουλία Ασφαλεία. Οπότε η Ευρώπη δεν μπορεί να καταφέρει, η Ένωση δεν καταφέρει να μιλήσει μια φωνή στη Σουηδική Προεδρία η απάντησή μου είναι είμαστε πολύ απεσιόδοξοι ώστε θα πετύχουμε κάτι. Δεν σας υπόσχομαι τίποτα. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα υποστηρίξουμε το ICC, δηλαδή και εκεί είναι δύσκολο θέμα η ειρηνευτική διαδικασία, Σουδάν, Νταρφούρ, το θέμα Βορρά-Νότου, η απογραφή, οι εκλογές που θα γίνουν στη χώρα αυτή Λευκορωσία. Θα συναντήσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών την Τρίτη. Τα σημεία αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη. Είχαμε ήδη, έχουμε ξεκινήσει μια, η Επίτροπος Βάλτερ ήταν εκεί, πρόεδρος Λουκασέγκο, και αυτός παίρνει μέρος στη συζήτηση, σίγουρα η φωνή μας θα είναι σαφής στο θέμα αυτό. Μέση Ανατολή, Συρία, ο Υφυπουργό Σουηδό ήταν εκεί πρόσφατα στη Δαμασκό για συζήτηση. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η δυνατότητα που υπάρχει να συμβάλλει στην ειρηνευτική διαδικασία για το Λίβανο, για το Ισραήλ, ίσως λίγο λιγότερο επιρροή στο Ιράν, παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες. Το έχουμε και αυτό. Το πιο αποτελεσματικό εργαλείο είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. έχουμε το πιο ισχυρό εργαλείο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ό,τι συμβαίνει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και δεν είναι μόνο για τα χώρε μέλη τη Ένωση, είναι και για τη Ρωσία, Φερρυπίν. Υπήρξα πρόεδρο τη Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου τη Ευρώπη για ένα διάστημα. Μετά η Ισπανία, μετά η Σλοβανία και όλοι συνεργαζόμαστε προκειμένου να ενισχυθούν αυτοί οι μηχανισμοί. Πρέπει να υποστηρίζετε το δικαστήριο στη δράση του και όλοι να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του. Ούτε και η Σουηδία είναι άγγελος. Υπήρξαν και περιπτώσεις που αφορούσαν τη Σουηδία, ότι έκανε, διέπρεξε παραβάσεις, παραβιάσεις όχι ιδιαίτερα σοβαρές, αλλά και οι ελάσσονες παραβιάσεις είναι παραβιάσεις και για τη Σουηδία. Και χάσαμε περιπτώσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό το θεωρώ θετικό. Διότι όταν πάω σε άλλες χώρες μπορώ να πω, δεν κάνουμε μόνο κήρυγμα. Αυτά οι αποφάσεις και τα όργανα αυτά παίρνουν αποφάσεις και για μας. Και πρέπει να σεβόμαστε και να εφαρμόζουμε αυτές τις αποφάσεις. Αναφέρθηκε η Συμφωνία της Άγκυρας, το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Υποθέτω εννοείστε το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Ναι, το είπα και πριν για τα πορίσματα του Συμβουλίου. Δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα στοιχεία και πρέπει όλα αυτά να τηρούνται. Νομίζω απάντησε στο σημείο αυτό πριν. Ονδούρα. Νομίζω κάναμε το σωστό. Υποστηρίζουμε τον πρόεδρο Αρίας και τις προσπαθίες του. Έχει μια έμεση εντολή από την Οργάνωση Αμερικανικών Κρατών και γιατί έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, είναι, έχει ένα πολύ άψογο παρελθόν και για φιλοσοφικούς γενικούς λόγους. Όπως ελπίζω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι πιο αποτελεσματικά στο μέλλον για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της, και της δημοκρατίας στην Ευρώπη, έτσι πρέπει να ενθαρρύνουμε και τον οργάνωση των Αμερικανικών κρατών, την οργάνωση για των εθνών των κρατών της Νότιο-Ανατολικής Ασίας ή της Αφρικής να παίρνουν τις αποφάσεις, να κάνουν την προσπάθεια να προσπαθήσουν να επιλύσουν τα προβλήματα των χωρών τους μόνοι τους. Οπότε θα έλεγα όχι εμείς να, παρέ, να παρέμβουμε αμέσως, να υποστηρίξουμε αυτές τις οργανώσεις να αναζητήσουν λύση. Αν αυτό αποτύχει, τότε θα έχουμε δύσκολες αποφάσεις τι θα κάνουμε με τις εμπορικές συμφωνίες και διάφορες άλλες συμφωνίες αλλά αυτό είναι κάπως διαφορετικό. Τέλος για την αλλαγή του κλίματος. Δεν το σχολίασα καθόλου. Θα μεταφέρω το θέμα αυτό, το σχόλιο, σε αυτούς που ασχολούνται ιδιαίτερα με το θέμα. Γεωργία. Ήμουν σε αποστολή 24 ώρες για να δω πώς λειτουργούν τα πράγματα επί τόπου. Κοιτάξτε, για τη διαχείριση των κρίσεων τα δύο τελευταία χρόνια αυτό που κάναμε απέδειξε σε σχέση με το παρελθόν ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Έχουμε επιτυχής δύσκολες αποστολές. Είχαμε αποστολή στο Τσάντ και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ σκληρή εντολή, δύσκολη κατάσταση και πετύχαμε. υπό έναν Ιρλανδό στρατηγό με Σουηδούς, Βέλγους, Ρουμάνους, ένα σωρό στρατιώτες. Αποδείξαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή πολιτική και στρατιωτική. Κανένα άλλο δεν μπορεί να το κάνει. Ούτε τα Ηνωμένα Έθνη κανένα δεν μπορεί να το κάνει. Φέραμε σε πέρα το έργο και μετά το παραδώσαμε στα Ηνωμένα Έθνη. Μετά έχουμε την αποστολή τη Αταλάντη. Κάτι που δεν μπορούσε κανεί να το δινοηθεί πριν από μερικά χρόνια. Κι όμω απέδωσε. Σημαντική συμβολή η δική μα και αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα πέραν αυτού που πολλοί θα θεωρούσαν ότι ήταν δυνατό πριν από μερικά χρόνια. Και όλα αυτά γίνανε μέσα σε πολύ λίγες μέρες, 10 μέρες, 14 μέρες. Νομίζω ότι η συμβολή προς σταθεροποίηση μιας πολλής ε, με, με, ε, κατάσταση η οποία μεταβάλλεται πολύ γρήγορα στην Απχαζία, παραδείγματο χάρη, η, επιτυχία ήταν σαφής. Βέβαια, η εντολή είναι να καλύψουν όλη την επικράτεια της Γεωργίας. Και παίρνουν στα σοβαρά αυτή την εντολή, περιπολούν σε όλη τη Γεωργία, όπου μπορούν να, να κάνουν αυτές τις περιπολίες. Ξέρουμε ότι όλες οι, οι διεθνείς οργανώσεις δεν τους επιτρέπονται μετά τον πόλεμο να μπουν στην Απχαζία και την Νότια Οσετία. Δεν μας αρέσει αυτό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι δυνατότητα έχουμε να υποστηρίξουμε τις ανθρωπιστικές δράσεις των ΟΕΕ Εθνών και λοιπά στην Απχαζία για να προστατευτούν αυτοί που χρειάζονται προστασία και επιμένουμε στα δικαιώματα του ΕΜΕΦ, το δικαίωμα της ΟΕΕΦ να παρακολουθεί την κατάσταση στην Οσετία και και στην, στην Απχασία και την Νότια Οσετία. Αυτό δεν λέω ότι θα το πετύχουμε πολύ σύντομα, αλλά μιλάμε για πολιτική, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, ακόμα και αν δεν πετυχαίνει βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντική γιατί είναι και θέμα αρχή και αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον. Η EMM λοιπόν έχει πολύ σταθεροποιητικό ρόλο στη Γεωργία, παίρνουμε εντολή από το Συμβούλιο να παραταθεί και αυτό υιοθετεί μια πολιτική αρχών που είναι σημαντική για την μακρόπνοη επίλυση διαφορών. Αυτό αφορά τον Κάφκασο και άλλες περιοχές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό για την πλήρη αυτή ε, παρουσίαση και απαντήσεις. Είναι πρόδρομος, φαντάζομαι, μιας συνεργασίας που θα συνεχιστεί στους επόμενους μήνες υπό την ηγεσία της Σουηδικής Προεδρίας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Σας ευχαριστούμε για μια φορά ακόμη και Υπουργέ. Ευχαριστώ όλους σας. Μετά τον αποχαιρετισμό με τον Υπουργό διακόπτουμε για μερικά λεπτά και μετά συνεχίζουμε. Uh, Συνεχίζουμε με ανακοινώσει για τα επόμενα σημεία τη ημερήσιας διάταξη. Έχετε πάρει δύο φακέλου που έχει ετοιμάσει η γραμματεία. Ο πρώτο μόνο στα αγγλικά. δραστηριότητε τη ε, επιτροπή στην προηγούμενη πενταετία. Το δεύτερο, InfoKit, δεύτερος φάκελος, σας πληροφορεί για τα πεδία δράσης της Επιτροπής Εξωτερικών. Έχουμε το πλαίσιο και τις επόμενες, αν θέλετε, τις επόμενες φάσεις της δουλειάς μας. Μόνο στα αγγλικά. Αρχές Σεπτεμβρίου θα το έχουμε σε όλες τις γλώσσες. για να ξέρετε τι σας περιμένει. Το πρωί συνεδρίασε το Προεδρείο και αποφάσισε να δώσουμε στον συνάδελφο Πέτερλε την έκθεση για την εταιρική σχέση με το Τατζικιστάν. Επίσης, η συνάδελφος Νέιτς Βίτενμπροικ πήρε την έκθεση για τον προϋπολογισμό 2010. Και έχουμε και το χρονοδιάγραμμα των ε, προσεχών συνεδριάσεών μας. Περνάμε στο επόμενο σημείο λοιπόν, που είναι η έκθεση για τον προπολογισμό 2010 της Επιτροπής Εξωτερικών. Η συνάδελφος Νέιτς. Uh, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη σας ότι εγώ είμαι εισηγητής αυτής της γνωμοδότησης, εισηγήτρια, διαδεχόμενη τη συνάδελφο που δεν επανεξελέγει και γι' αυτό ανέλαβα εγώ το έργο της. Μου ζητήθηκε λοιπόν να το αναλάβω εγώ. Το κάνω, παρόλο που ο προπολογισμό δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω. Έχουμε λοιπόν ήδη κυκλοφορήσει σήμερα και ευχαριστώ τη γραμματεία που το έχει κάνει και τους δικούς μου βοηθούς για τη βοηθειά τους. Κυκλοφορήσαμε λοιπόν δύο έγγραφα ένα σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής μας για τον Γενικό Προϋπολογισμό, που είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προϋπολογισμών και ένα έγγραφο εργασίας με διάφορες παρατηρήσεις που σας υποβάλλω εγώ. Εκεί υπάρχουν και διάφορα διάφορες προτάσεις τροπολογιών που σας υποβάλλω. Εννοείται ότι πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνουμε, κατά πόσο θέλετε να καταθέσουμε αυτές τις τροπολογίες ή αν έχετε κι άλλες, γιατί αν δεν απατώμε η προθεσμία για κατάσταση τροπολογιών είναι 25 Αυγούστου. Μέχρι τότε λοιπόν μπορείτε εσείς να καταθέσετε τροπολογίες στη γνωμοδότηση αυτή. Ποιες είναι οι κύριες πτυχές λοιπόν τώρα του τμήματος αυτού του σχεδίου προϋπολογισμού. Ο τίτλος 4. Αυτό το οποίο εκπλήσει είναι ότι γενικά δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια εδώ. Όπως ξέρουμε δεν είναι η πρώτη χρονιά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Καφέ άλλο. Και τόσο η Επιτροπή, αλλά ακόμα περισσότερο το Συμβούλιο, το κάνουν γιατί ξέρουν ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί να προκύψουν διάφορες επίγουσες καταστάσεις και έτσι οι υπηρεσίες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν χρήματα. Θα ανοίξουν όλα τα ζυρτάρια, τα τελευταία ό,τι έχει μείνει θα φροντίσουν να τα βάλουν μαζί για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες. Εμείς όμως δεν συμφωνούμε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος μακροπρόθεσμα για να προετοιμάζουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τρόπος για να καλύψουμε τις πολιτικές μας. Τώρα, η μείωση στις υποχρεώσεις εξηγείται εν μέρη από την χρηματοδότηση του μέσου διευκόλυνσης σύντησης που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Food Facility Instrument και που χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό του 2009. 47% από ένα εκατομμύριο. Ένα δις, συγγνώμη. Από ένα δις. Το υπόλοιπο είναι από τον προπολογισμό του 2010. Αυτό το οποίο επίσης μας εκπλήσει και εγώ βρίσκω απαράδεκτο είναι η συνολικά μία ρεαλιστική μείωση της χρηματοδότησης για την Παλαιστίνη. Πρέπει να επιμείνουμε ότι η κύρια διαδικασία επί του προϋπολογισμού αποτελεί και τη βάση εργασίας μας. Δεν είναι σοβαρό να μειώνουμε το ποσό. Δεν είναι ρεαλιστικό. Γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα χρειαστεί αύξηση των ποσών και θα πρέπει κάπου να τα βρούμε αυτά τα χρήματα. Κάπου αλλού. Άλλη παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το συνολικό ποσό για τις πληρωμές είναι μικρότερο από τις προηγούμενες χρονιές επειδή η, η υποχρέωση τα περίφημα ΡΑΛ rest alikide έχουν μειωθεί ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός εφαρμογής των πολιτικών έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Ελπίζω να είναι όντως έτσι. Τώρα υπάρχουν 220,8 εκατομμύρια ευρώ, 2,8 δηλαδή του τίτλου 4, έχει μπει Ε, έχει παγώσει και είναι πέρα από το σύνολο του προπολογισμού. Είναι ένα περιθώριο ελιγμών, θα μπορούσαμε να πούμε, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας συγχρόνως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να αυξήσει εφόσον χρειάζονται υποχρεώσεις για την Παλαιστίνη. Και θα χρειαστεί και να αυξήσει τα ποσά και για την Κούβα, τη Γεωργία, το Κωσυφοπαίδιο και ενδεχομένω και για την επανένωση στην Κύπρο και για πρωτοβουλίες στα πλαίσια της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Όλα αυτά πρέπει να χρηματοδοτούν από αυτό το περιθώριο. Καταλαβαίνετε ότι ήδη έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσό, οπότε ειλικρινά δεν είναι ρεαλιστικό να το παρουσιάζουμε σαν περιθώριο. Τώρα, οτιδήποτε επιπλέον κονδύλια για άλλες προτεραιότητες ή για άλλα πρόβλεπτα γεγονότα, μια φυσική καταστροφή, ένας θεός ξέρει τι, μέσα στο 2010 θα μας φέρει αντιμέτωπους με τεράστιες δυσκολίες προκειμένου να βρούμε χρήματα. Τώρα το Συμβούλιο έχει μειώσει τις υποχρεώσεις για το κεφάλαιο 4 κατά 89,11 εκατομμύρια και έχει μειώσει τις πληρωμές κατά 259,47 εκατομμύρια αυξάνοντας το περιθώριο που μένει για την Επιτροπή σε 309,90 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 220,8 είχε βάλει και το Συμβούλιο αύξησε το ποσό στα 309,90 εκατομμύρια. Τώρα το αρχικό προσχέδιο μιλούσε για 7,9 σε σύγκριση με 8,1 εκατομμύρια που είχαμε πέρυσι. Μείωση λοιπόν 2,3%. Και οι πληρωμές που προτείνονται σημαίνει μείωση 7,9%. Η συνολική χρηματοδότηση για το μέσο γυτνίασης είναι λίγο χαμηλότερο από ό,τι το 2009 είναι μια μείωση που εξηγείται από μη ρεαλιστικές χαμηλές υποχρεώσεις και πληρωμές για την Παλαιστίνη, αλλά αυτά σας τα είπα ήδη. Οι υποχρεώσεις για το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως επίσης και οι υποχρεώσεις και οι πληρωμές για το Μέσο για την προενταξιακή διαδικασία, είναι όπως και το 2009. Όμως πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι για το 2010 100 εκατομμύρια ευρώ πάνε από την πολιτική γετνίασης και την προενταξιακή διαδικασία και από ένα άλλο μέσο για να χρηματοδοτηθεί το Food Facility Instrument, η σύντηση με πιστοφή το 2011 κλπ. Να λοιπόν ένα παράδειγμα τι γίνεται όταν οι προβλέψεις μας δεν είναι ρεαλιστικές. Τελικά τι γίνεται. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς συμβαίνουν πράγματα, όπως για παράδειγμα ε, δανειζόμαστε χρήματα από άλλες πηγές, τα οποία πρέπει να επιστρέψουμε αργότερα. Οπότε είσαστε αντιμέτωποι με ποσά και ένα προπολογισμό που σε ορισμένε πτυχέ τουλάχιστον έχει σχέση με την πραγματικότητα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το 2010. Για μένα αυτή δεν είναι μια καλή βάση για να ετοιμάζει κανείς ένα προπολογισμό. Το Συμβούλιο επίσης πρότεινε να μειώσει και τις διοικητικές δαπάνες σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορες γραμμές. Εδώ βέβαια μπορώ να φανταστώ γιατί το κάνει αυτό το Συμβούλιο. Θεωρεί ότι να, αυτό είναι εύκολο. Βλέπετε μια γραμμή διοικητικές δαπάνες, το διαγράφετε, λέτε. Α, ας κάνουν χωρίς. Ναι, αλλά συγχρόνως εμείς θέλουμε οι διάφορες πολιτικές μας να φέρονται σε πέρας ικανοποιητικά, σωστά, αποτελεσματικά. Και θέλουμε αυτό να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν όμως δεν έχετε αρκετό προσωπικό δικητικό για να το κάνει, ε, πώς θα γίνει. Οπότε αν μειώνετε τις διοικητικές δαπάνες υπερβολικά, ουσιαστικά παγιδεύετε την ίδια σας την πολιτική. Για άλλη μια φορά λέω ότι αυτός δεν είναι σωστός τρόπος για να φτιάχνουμε τον προπολογισμό. Τέλος, προτείνω μια τροπολογία που προσθέτει χρήματα στη γραμμή 02 για τη στρατηγική μας στην Βαλτική θάλασσα. Δεν έχει χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση εδώ. Τώρα οι συνάδελφοι της περιοχής προτείνουν να προσθέσουμε 20 εκατομμύρια στην γραμμή του προπολογισμού, που εγώ θεωρώ ότι ίσως είναι υπερβολικά γενναιόδωρο. Οπότε θα δούμε το Σεπτέμβριο τι τελικά θα κάνουμε με το ποσό. Συνάδελφοι, αυτές είναι οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω και που προτείνω ώστε να βάλουμε λίγο ρεαλισμό στην πρόταση αυτή για τον προϋπολογισμό. Τόσο για τις υποχρεώσεις όσο και για τις πληρωμές. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω όλα όσα όπως μας είπε η συνάδελφος. Τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί συχνά με τον προπολογισμό γιατί ήμουν και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Η γενική μου εντύπωση είναι πως ασχολούμαστε με τα νούμερα στις επιτροπές και εγκρίνεται μετά από διαπραγματεύσεις ο προϋπολογισμός, αλλά κατ' ουσίαν μιλάμε για μία φωτογραφία, μία μόνο χρονική στιγμή και μετά αλλάζουν τα νούμερα συνεχώς και έρχονται τροπολογίες, ε, εκκλήσεις κομισιών να γίνουν αλλαγές. Ε, Και αυτό ισχύει κυρίως για τον τίτλο 4, στις εξωτερικές υποθέσεις. Έχουμε αυτή την χρόνια υποχρηματοδότηση και συγκεκριμένα στον τομέα της Παλαιστίνης ε, επί σειρά ετών έχουμε ξεφύγει όσον αφορά την εφαρμογή του προϋπολογισμού και θα πρέπει να γίνει επιτέλους κάπως πιο ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός. Η Κομισιόν να το δει πιο μακροχρόνια και να μην είναι συνεχώς τόσο μη ρεαλιστικά αυτά τα, τα νούμερα και κάθε δύο εβδομάδες να υπάρχει τροποποιητική επιστολή από τους επιτρόπους που μας ε, ζητάει νέα κονδύλια λόγω της κατάστασης. Οπότε η κριτική και στο συγκεκριμένο σημείο της Παλαιστίνης με βρίσκει σύμφωνο. Επίσης στο σημείο 5 των προτάσεων σύμφωνο όπου ασκούμε κριτική στη μείωση των κονδυλίων στον Ευρωπαϊκό Μέσο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το μέσο αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα και θα αναφερθώ εδώ στο Ιράν. Δεν ναι, θέλουμε βλέπουμε τα χειρότερα σενάρια να επιβεβαιώνονται απ' έξω, μπορούμε να τα αλλάξουμε από μέσα, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο. Γιατί λέμε ναι αυτό είναι το μέσο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρίς την ε, σύμφωνη γνώμη των ε, εμπλεκομένων ε, κυβερνήσεων. Π.χ. υπάρχουν στο Ιράν δικηγόροι που υπερασπίζουν ανθρώπους Χωρί σύμφωνη γνώμη τη ε, Νομίζω γι' αυτό υπάρχει αυτό το, το μέσο. Και καλό θα ήταν να μην περιοριστεί το ποσό που υπάρχει εδώ πέρα. Αυτά. Πιθανώς να καταθέσω και κάποιες ε, τροπολογίες για να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βασικά συμφωνώ με την εισηγήτρια, ιδιαίτερα με τις παρατηρήσεις που έκανε για την υποχρηματοδότηση στην κατηγορία αυτή του προπολογισμού. Και όσον αφορά επίσης το περιθώριο, το οποίο βασικά αφήνει χωρίς περιθώριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αρχές επί του προπολογισμού για να αποφασίζουν για νέες περιπτώσεις που προκύπτουν και που χρειάζονται χρηματοδότηση. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τον ενισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές επίπεδο με ένα τέτοιο προπολογισμό, γιατί ο προπολογισμό όντω αποτελεί μια φωτογραφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πώ ανταποκρίνεται αυτό στι προσδοκίε μα όταν μειώνουμε τα κονδύλια. Το Food Facility δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις που έχουν άλλο προορισμό. Στις χώρες μας και στη δικιά μου έγιναν προσπάθειες για να ανταποκριθούμε στις επιστηστικές ανάγκες με άλλα κονδύλια. Μα δεν είναι δυνατόν ε, να τα παίρνουμε από το ένα χέρι για να τα δίνουμε στο άλλο. Στο προσχέδιο προϋπολογισμού υπάρχουν πολλά υπόμνηση όσον αφορά τη Λατινική Αμερική. Εδώ θα ήθελα να μας το εξηγήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Λόζινγκ τώρα. Ναι, μιλήσαμε για τη χρόνια υποχρηματοδότηση του προϋπολογισμού και στην έκθεση της, ε, του Λάσλο Σόγεν και στην έκθεση της κυρίας Νέιτς λέγεται πως πρέπει να λάβουμε πολλές αποφάσεις χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πράγματι πρέπει να γίνουν αλλαγές στον προϋπολογισμό. Η τα αυξημένα κονδύλια που χρειάζονται για την εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να επενδυθούν σε στρατιωτικές δραστηριότητες αλλά στην καταπολέμηση της στόχιας στις αναψώμενες χώρες, οικολογική μεταστροφή, δικαιώματα των γυναικών κτλ. Και να αναλάβει το κόστος σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 για μέτρα στρατιωτικά κτλ. Είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται να το πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε εάν πραγματικά απαιτούνται όλα αυτά τα έξοδα. Πρέπει να εξεταστούν κάποια πράγματα όπως π.χ. το σύστημα Γαλιλαίο ή το μέσο για την ειρήνη. Π.χ. πόσα λεφτά πήγανε το 2010 για τον Γαλιλαίο που έφυγαν από τη γεωργική πολιτική. Επίσης η απαγόρευση της λεγόμενης ε, παράλληλης ε, χρηματοδότησης και το μέσο υποστήριξης της ε, ειρήνης, το οποίο υποτίθεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για άμεση καταπολέμηση της στόχης. Δεν θα αναφέρω και άλλα παραδείγματα ε, για τα οποία θεωρώ πως γίνεται στρατιωτική χρήση των ε, κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως π.χ. ο Μηχανισμός Αθηνά και λοιποί. θεωρώ πως ε, εάν πάνε τα χρήματα αυτά μόνο σε πολιτικές μη στρατιωτικές χρήσεις θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια χαρακτηριστική κατάσταση όσον αφορά τον προπολογισμό και η συγκήτρια της Επιτροπής μας μας παρουσιάζει κάποια στοιχεία πάρα πολύ συγκεκριμένα με συμβιβασμού στις υποχρώσεις και στις πληρωμές. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κ. Γκάλερ και θα συνεχίσω από εκεί. Χρειάζεται διευκρίνηση επί της διαδικασίας. Έχουμε δύο έγγραφα. Ένα σχέδιο γνωμοδότησης που σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη μπορούμε μέχρι τις 25 Αυγούστου να τροποποιήσουμε και ένα έγγραφο εργασία το οποίο έχει να κάνει με την παρουσίαση τροπολογιών από την ίδια την εισηγήτρια της Επιτροπής μας. Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να τροποποιήσουν, φαντάζομαι, το σχέδιο γνωμοδότησης και θα υπάρξει προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών στα νούμερα, στα ποσά που είναι στις διάφορες γραμμές. Πολύ σωστά ο κύριος Γκάλερ παρουσίασε τη θέση της πολιτικής μας ομάδος, δηλαδή τα επιχειρήματα που ανέφερε και η συγγύτρια. Θέλω να προσθέσω, και το είπε και ο Υπουργό σήμερα, πόσο μεγάλη σημασία έχει η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, θα έχουμε μία ανακοίνωση από τους Υπουργούς που θα μιλάει για τις εξωτερικές δράσεις εφόσον εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Οπότε από εκεί και πέρα θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη δημοσιονομική για να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα σχόλια πάντως της κυρίας Νέιρς είναι σωστά όσον αφορά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Παλαιστίνη ειδικότερα. Πολύ σωστά επίσης είναι αυτά που λέει για το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γι' αυτό το σημείο σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον συνάδελφο Μπροκ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Τσετσενία μετά από διάφορες επισκέψεις. Καλό θα ήταν, πιστεύω, να μελετήσουμε, να δούμε μήπως μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες με στόχο να ενισχυθεί η δράση στην περιοχή υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μια που ξέρουμε ότι τελευταία έγιναν και διάφορες δολοφονίες εκεί. Γενικά μιλώντας, αυτά ήταν τα σχόλια που είχα να κάνω πρόεδρε και θέλω διευκρίνηση για την διαδικασία, όχι όσον αφορά την γνωμοδότηση, που από ό,τι κατάλαβα εδώ μπορούμε μέχρι τις 25 του μηνός να υποβάλουμε τροπολογίες, αλλά για τις συγκεκριμένες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τις δημοσιονομικές γραμμές, με τις γραμμές των προπολογισμών. Εκεί θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με τις τροπολογίες. Θα απαντήσω αφού συζητήσω με τη γραμματεία. Μέσα στον Αύγουστο θα υποβληθούν τροπολογίες στην έκθεση συναδέλφου Νέιτς και για το σύνολο του προπολογισμού 2010, αλλά τη συγκεκριμένη ημερομηνία 25 Αυγούστου σα τη δίνω ω τελική προθεσμία με ενδεχόμενε προσαρμογές αυτό θα το πω στο τέλος τη συνεδρίαση. προκειμένου να ψηφίσουμε την έκθεση στις 2 Σεπτεμβρίου. Χάουτολα. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων σας δηλώνω ότι μας ευχαριστεί η γνωμοδότηση της κυρίας Νέιτς και ιδιαίτερα για την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χαίρομαι για το ότι τονίζει το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένας πολύ αποτελεσματικό καλός τρόπος να ξοδεύουμε τα χρήματα που διαθέτουμε. Και όπως λέει η κυρία Νέτς, θα πρέπει να ζητήσουμε όλα αυτά να χρησιμοποιηθούν με συγκεκριμένους στόχους, αλλά και με ευέλικτο ταυτόχρονο τρόπο. Θα υποβάλουμε ορισμένες τροπολογίες, όπου θα τονίζουμε τη χρησιμότητα αυτού του μέσου για το Βόρειο Κάφκασο, όπου η κοινωνία των πολιτών περνάει δύσκολες στιγμές. Πρόεδρος. Αντρικίνεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Νέιτς για την γνωμοδότηση. Η κατηγορία 4 του προπολογισμού συνήθως ε, έχει ανεπαρκή κονδύλια. Φιλοδοξία μας είναι να ενισχυθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ένωσης προς το εξωτερικό. Και θα ήθελα να αναφερθώ και την ε, στρατηγική για τη Βαλτική, που είναι μια από τις προτεραιότητες της Σουηδίας. Το ακούσαμε σήμερα από τον Υπουργό Εξωτερικών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να ενισχύσει την στρατηγική αυτή τον Οκτώβριο, από ό,τι ακούμε. Και μετά θα αρχίσει η εφαρμογή της. Εμείς συντάσσουμε εδώ το πρόγραμμα δράσης. Συμφωνώ με την γνώμη της εισηγήτριας. 20 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω για την εφαρμογή της στρατηγικής για το 2010. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Τελειώσαν οι παρεμβάσεις των συναδέλφων. Τώρα οι κύριοι Γκέρι Μίλλερ και Αντρέα Ηλιής της Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Η συγγήτρια, η συγγήτρια, θέλετε να μιλήσετε τώρα, κύριε Νέιτς. Πολύ σύντομα στο σχέδιο γνωμοδότηση σελίδα 6 στην τελευταία σειρά λέει συνεχιζόμενη οικονομική βοήθεια προς του τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η λέξη κυπριακή έφυγε. Χάθηκε μας την υπολογιστή πρόεδρος. Όπως είπε ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο διάβολος κρύβεται πίσω από τις λεπτομέρειες. Λεπτομέρεια ήταν αυτή. Κομισιόν ο κύριος Μίλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Γκάρι Μιλίν, επικεφαλή οικονομική μονάδα στη Γενική Διεύθυνση για τι Εξωτερικέ Σχέσει. Θα ήθελα να πω στου νέου ευρωβουλευτέ ποιο είναι ο ρόλο τη Κομισιόν. Διευκολυντικό είναι. Είμαστε στη διάθεση των βουλευτών να σας βοηθήσουμε στην δουλειά αυτή για τον προπολογισμό που δεν είναι εύκολη και θα πρέπει καταρχήν να συγχαρούμε την κυρία Νέης που της δόθηκε αυτό το δύσκολο έργο. Είμαστε στη διάθεσή σας, στη διάθεσή της και εμείς και όλη η υπηρεσία μας για την επεξεργασία της γνωμοδότησης αυτής, την εκπόνησή της. Ο Γενικός Διευθυντής μου και η Επιτροπή ε, στις περισσότερες περιπτώσεις βρισκόμαστε, λειτουργούμε στο ίδιο μήκο κύματο. Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τη Γενική Διεύθυνση για τη Διεύρυνση, Θέλω να σα πω γιατί είναι υπεύθυνη η δική μου γενική διεύθυνση για τι εξωτερικέ σχέσει και τον προγραμματισμό των μέσων, το μέσο γειτονία, το, το αναπτυξιακό μέσο, ο προπολογισμό για τι εξωτερικέ δράσει, ε, μέσω διαχείριση κρίσεων, CFSP, και το μέσο σταθερότητας. Αυτά είναι τις δικές μας αρμοδιότητες και ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση για τη Διάβηση θα μιλήσει για τα... τις δικές του υποχρεώσεις. Ακούσαμε ότι υπάρχει ανεπάρκεια στα κονδύλια όσον αφορά τα... τις εξωτερικές δράσεις. Αυτό το λέει στο κείμενό της η συγγήτρια. Κάθε χρόνο εμφανίζεται το θέμα αυτό η Κομισιόν θεωρεί ότι στις προτάσεις μας για τον προπολογισμό για το 2010 κάνουμε σωστές εκτιμήσεις για τα προγράμματα που υπάρχει βεβαιότητα δαπάνης. Έπρεπε να κάνουμε την εκτίμηση το Μάιο τι θα ξεδέψουμε για τον επόμενο χρόνο. Είναι δύσκολο το έργο αυτό. Αυτό που γίνεται και είναι φυσιολογική διαδικασία, λέμε, προς το τέλος της χρονιάς μπορούμε να επανέλθουμε και να τροπολογήσουμε την πρόταση. Αυτό το επιτρέπει η δημοσιονομική διαδικασία. Ήθως ήταν κάπως ατυχέ αυτό το ότι έγινε τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή είχαμε ένα σωρό προκλήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι τις περισσότερε φορέ να αναθεωρήσουμε μερικέ από τι προτάσει μα. Γιατί οριστικοποιούνται τα προγράμματά μα προ το τέλο του χρόνου, μέσα όπω τρέχει η χρονιά. Ίσως το πιο σημαντικό θέμα σε όλα αυτά είναι η Παλαιστίνη. Και εμείς συμφωνούμε με αυτό. Χρήσιμο για μας θα είναι να επανέλθουμε με άλλη πρόταση αργότερα, αφού θα έχουμε αξιολογήσει και τις προσπάθειες των άλλων δωρητών για την Παλαιστίνη. Το Σεπτέμβριο, στις αρχές του μηνός, η Κομισιόν θα εγκρίνει τροπολογία, τροποποιητική επιστολή τη λέμε, στο σχέδιο αυτό, όπου η Παλαιστίνη θα υπάρχει μέσα. Ένα άλλο αρκετά σημαντικό θέμα επίσης, και θα επανέλθω σε αυτό, είναι η διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο τέλος του χρόνου. Είναι προτεραιότητα για τον πρόεδρο Μπαρόσο. Το αν έχουμε ή όχι επαρκή κονδύλια, αν υπάρχουν νέες ανάγκες, νέες προτεραιότητες, θα βρούμε λύση. Οι παλιοί βουλευτέ θυμώνται ότι βρήκαμε λύση για την εταιρική σχέση με την Ανατολή, με, με το μέσον για την ε, επιστηστική βοήθεια. Όλα αυτά τα προβλέπει η δημοσιονομική διαδικασία. Η κατάσταση λοιπόν δεν πρέπει να την περιγράφουμε με μελανά χρώματα. Αναφέρθηκε ένα ερώτημα για το περιθώριο ελιγμών από το 2011 και μετά. 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο. Η Κομισιόν και ιδιαίτερα σε θέματα της οικογένειας του Ρέλεξ θα προβληματιστεί. Τα σημειώσαμε πάντως τα σχόλια αυτά για την αναθεώρηση του προπολογισμού. Είναι μια αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και είπαμε τα τρία όργανα ότι θα επανέλθουμε σε έναν ενδιάμεσο χρόνο για αναθεώρηση. Θα γίνει μια ενδιάμεση αναθεώρηση. Θέλει είναι μια σημαντική ευκαιρία αυτή η αναθεώρηση χρονικά. Τμήμα της περσινής συμφωνίας για το Food Facility, το μέσο διατροφής, η Κομισιόν συμφώνησε να κάνει μια ειδική αξιολόγηση απολογισμό στον προπολογισμό για εξωτερικές δράσεις. Τον Σεπτέμβριο θα το κάνουμε αυτό με την τροπολογητική, τροποποιητική επιστολή μας. Στο κεφάλαιο 4 και τι εξελίξει θα έχει το περιθώριο ελιγμών από σήμερα μέχρι το 2013. Τώρα απαντήσει σε συγκεκριμένα σχόλια της εισηγήτρες. η Κομισιόν επικροτεί τις προσπάθειες της εισηγήτριας να αποκατασταθεί η αρχική πρόταση της Κομισιόν. Είναι ένα είδος λοιπόν κλασική. Η Κομισιόν κάνει προτάσεις, το Συμβούλιο κάνει την πρώτη κίνηση, εγκρίνει το σχέδιο προπολογισμού, πριν από μια εβδομάδα γίνει αυτό, με περικοπές, έρχεται στο Κοινοβούλιο και το Βούλιο κρίνει αν δέχεται αυτές τις περικοπές ή όχι. Βέβαια η Κομισιόν δεν τις θεωρεί αποδεκτές τις περικοπές αυτές. Τώρα αν η κυρία Νέιτς θέλει να αποκαταστήσει ορισμένα κονδύλια θα μας βρει σύμφωνος. Και όπως είπε η κυρία Νέιτς, πρέπει να αποκατασταθεί το επίπεδο ε, κονδυλίων ε, δεσμεύσεων, ιδιαίτερα στο DCI, και πιο συγκεκριμένα για τον προπολογισμό για την πολιτική πληροφόρηση. Επίσης συμφωνούμε να αποκαταστεί το αρχικό ποσό όσον αφορά τις ε, πληρωμές. Είναι τα χρήματα που πραγματικά μπορούμε να δαπανίσουμε. Η πρόταση του Συμβουλίου στην κατηγορία 4 περιέκοψε 500 εκατομμύρια αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Το νέο όργανο RELEX αυτή τη στιγμή ε, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται με μια καλή ταχύτητα και επιταχύνεται κιόλα. Οποιαδήποτε λοιπόν περικοπή, ιδιαίτερα σε τέτοιο μέγεθο, θα επιβραδύνει την υλοποίηση των προγραμμάτων. Επίσης υποκριτούμε την υποστήριξη τη εισηγήτρια για τον διοικητικό προπολογισμό τελειώνουμε πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο είναι μια τροπολογία που προτείνει 20 εκατομμύρια για την στρατηγική της Βαλτικής. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να καταλάβουμε ποια είναι η πρόθεση της ηγήτριας εδώ. Αν είναι τροπολογία για λόγους περιφερειακής πολιτικής, η Κομισιόν θα έχει κάποιο πρόβλημα να χρηματοδοτήσει αυτό το, το, τη δράση στο 4, γιατί είναι για εξωτερικέ δράσει το 4. Πρέπει να μα εξηγήσει η συγκεκριτή τι εννοεί, ποια είναι η πρόθεσή τη, Επίση αναφέρονται τα πιλωτικά προγράμματα και συνεφείς δράσεις. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε για να καταλάβουμε πού έγκυται τα προβλήματα, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Ευχαριστώ από τη Γενική Διεύθυνση Ρελέξ και αν επιτρέπετε να πάρει το λόγο στην από την ε, Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση. Ευχαριστώ. Ανρή Λύς λέγομαι. Είμαι υπεύθυνο ε, της οικονομικής ε, αρρωγής και του συντονισμού στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Προεδρία που μας τον λόγο για να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας και να συγχαρώ βεβαίως και τους ε, κυρίους και τις κυρίες ε, βουλευτές ε, είτε πανεξελέγησαν είτε τώρα εξελέγησαν για πρώτη φορά και βεβαίως αναμένουμε να έχουμε μαζί σας μία επικοδομητική συνεργασία. Να συγχαρώ και την κυρία Νάις που απεδέχθη αυτή την ευθύνη και είχαμε συνεργαστεί και με τον προκατοχό σας και θα στηρίξουμε και στο μέλλον. Όσον αφορά την διεύρυνση, το τόνισε και ο κύριος Μπίλτ, πρέπει να στείλουμε το στο μήνυμα στις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες ε, την ε, στιγμή αυτή που αντιμετωπίζουμε μια οικονομική κρίση. Και ε, βεβαίω πρέπει να υπάρχει μια στήριξη, αλλά έχει κοπεί και ο προϋπολογισμός και ο επιχειρησιακός ε, και ο λοιπός για το μέσο. Να σας προλάβω εδώ πέρα έχουμε προβλέψει εμείς αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το πολυετές ενδεικτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα που υποβάλλουμε κάθε έτος και αποτελεί υποχρέωση της ε, Κομισιόν σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα αναφερθώ στις μειώσεις του υπερπολογισμού στις επιχειρησιακές γραμμές και μετά η συνάδελφος θα καλύψει τις διοικητικές γραμμές για, για μικρότερα ποσά αλλά εξίσου σημαντικά. Πρώτα απ' όλα να συμπενθυμίσω κάποια πράγματα για την δομή του προενταξιακού μέσου ε, μπορεί να το ξέρετε, ίσως όχι, έχει η οικονομική εταιρική σχέση πέντε τμήματα. Έχουμε για το κράτος δικαίου, τη δημόσια διοίκηση, καθώς και την προώθηση των καλών γειτονικών σχέσεων στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Αυτά ισχύουν για όλες τις χώρες. Μετά έχουμε τρία άλλα στοιχεία που δεν ισχύουν για όλες τις χώρες, αλλά αφορούν μόνο τις υποψήφιες χώρες και έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως ανεργία, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση, επένδυση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταφορές, περιβάλλον καθώς και αγροτική ανάπτυξη. Το Συμβούλιο πρότεινε ε, κάποιες περικοπές και ειδικά όσον αφορά τις ε, γειτονικές ε, χώρες, κάτι το οποίο κατά την απόψή μας θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο. Όλα, πρώτα απ' όλα τα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν, θεωρούσαμε πως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις ε, χώρες αυτές να στήσουν τις δομές για την αποκεντρωμένη διαχείριση κονδυλίων, κάτι το οποίο σημαίνει προετοιμασία και ελέγχους ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, και προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση πριν ξεκινήσει η εφαρμογή. Γι' αυτό κατανέμονται τα κονδύλια στα τρία τμήματα που σας ανέφερα. Γι' αυτό επίτηδες είχαν ε, χαμηλό ποσό στο 2008-2009 καθώς ξεκινούσε το νέο μέσο για να μπορέσουν να στήσουν τις δομές τα κράτη-μέλη αυτά για την εφαρμογή. Οι υποψήφιες χώρες επέδειξαν καλή πρόοδο στον τομέα αυτό και θα πρέπει να τους δοθεί το πράσινο φως στο τέλος του έτους πριν ξεκινήσει η εφαρμογή. Αν γίνει αποδεκτή ε, η πρόταση του Συμβουλίου σημαίνει πως δεν αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής επιπλέον. Θα δείξουμε πως δεν υπάρχει αλληλεγγύη κατά τη διάρκεια της οικονομικής ε, κρίσης, καθώς ε, κατ' ουσίαν μιλάμε για αυτά ακριβώς τα μέσα που θα βοηθήσουν τις χώρες αυτές να περιορίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης. Μια άλλη σημαντική πτυχή που τόνισε η κυρία Νάις ε, είναι η σημασία της πολυετούς προσέγγισης και του προγραμματισμού της βοηθείας αυτής. Εμείς προγραμματίζουμε ορίζοντα τριών ετών και μετά τα κονδύλια κατανέμονται με αιτήσιες δόσεις και μέχρι στιγμής ε, το ποστό είναι 100%. Οπότε το να μην σεβαστούμε τις κατανομές που έχουμε ορίσει στον πολιετή προγραμματισμό βεβαίω θα, θα έχει καταστροφικό αποτέλεσμα. Επίση υπήρχε εντύπωση πως ήταν χαμηλέ πληρωμές το 2009, αυτό είναι σωστό, αλλά πέρα από το ότι έχει μειωθεί έχουν μειωθεί οι καθυστερήσει. Ε, αυτό αντικατοπτρίζει το ότι αυξάνονται οι πληρωμέ σε το χρόνο, κάτι το οποίο είναι παρόμοιο με το τι συμβαίνει με τα διαρθρωτικά ταμεία εντό τη Ένωση. Τώρα να δώσω τον λόγο στην συνάδελφο για τις ε, πτυχές τις διοικητικές και μετά να δεχτούμε ερωτήσεις. Ήδη η συγκήτρια υπογράμμισε τη σημασία που έχει να έχουμε αρκετό προσωπικό, πολύ βασικό για να μπορούμε να αποδώσουμε με τον προπολογισμό που έχουμε. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε λοιπόν μία ελαφρά αύξηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2010. Όμως θα είναι πάρα πολύ μικρός. Ο λόγος είναι ότι η Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης ανέλαβε όλα τα σχετικά με την ανοικοδόμηση στα Βαλκάνια, οπότε εκεί χρειαζόταν περισσότερο κόσμο σε ολόκληρη τη χρονιά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε το κοσυβοπαίδιο. Αναφέρθηκε πολλές φορές στη συζήτηση πριν και εδώ χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό στην Πριστίνα. Είναι επίση πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε, όπω είπε και ο συνάδελφο πριν, ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή των προγραμμάτων που χρειαζόμαστε διαχειριστική δύναμη. Το διοικητικό σκέλος είναι χαμηλότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει αρχικά, 25% λιγότερο ήδη. Παρ' όλα αυτά, το Συμβούλιο μας ε, περιέκοψε και μας έβαλε με ένα προπολογισμό λιγότερο από εκείνο του 2009, που έτσι καλώς δεν έφτανε. Ελπίζω λοιπόν να καταλάβετε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες οι περικοπές αυτές υπονομεύουν τις δυνατότητες των αντιπροσωπιών να φέρουν σε πέρα τους ελέγχους εξάντε που χρειάζονται για την αποκεντρωμένη διαχείριση. Όμως θέτει και σε αμφισβήτηση τη δυνατότητα των αντιπροσωπιών να ασκήσουν τον έλεγχο και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε λοιπόν υγιή οικονομική διαχείριση και νομιμότητα όσον αφορά τις ε, οικονομικές συναλλαγές. Η Επιτροπή γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ξέρουμε ότι μιλάμε για τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Όμως σε μια στιγμή οικονομικής κρίσης ο ορθός έλεγχος και ορθή ε, εφαρμογή στην πράξη του προπολογισμού είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Γι' αυτό και ζητάμε από εσά, από την Επιτροπή σα, να μα δώσετε τα κονδύλια που χρειαζόμαστε για να φέρουμε σε πέρα ε, το... τα καθήκοντά μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Κομισιόν και για το τελικό σχόλιο η συγγήτρια κυρία Νέιτς. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ε, σχολίασαν θετικά το σχέδιο. Πράγματι, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 25 Αυγούστου και προφανώς αφορά και το κείμενο και τους αριθμούς η προθεσμία. Μπορείτε να τροποποιήσετε και τους αριθμούς όχι μόνο αυτούς προτείνω εγώ να αλλάξουν, ε, οτιδήποτε αφορά τον τίτλο 4, εάν θεωρείτε χρήσιμο να, να κάνετε κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ευγενέστατα είπαν πως σε γενικές γραμμές συμφωνούν, οπότε το σημειώνω αυτό με ικανοποίηση. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Uh, and Madame de Bucci for uh, their comments uh, from the side of of the Commission, and I can assure them that after a a short summer break we will sit together and uh, to continue the work on on on the draft. Και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Θα συνεχίσουμε βεβαίως να εργαζόμαστε στο επί του σχεδίου αυτού. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. σα είπαμε πριν προθεσμοί για τροπολογίε 25 Αυγούστου. Πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεσή μα στι 2 Σεπτεμβρίου για να το στείλουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών μέχρι 9, για τις 9. τροπολογίες μόνο στα αγγλικά και στα γαλλικά. Δεν θα έχουμε χρόνο για μετάφραση. Και ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο για σήμερα, που είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν. Ο κύριος στον οποίο έχει δοθεί η εντολή να είναι εισηγητής. Πέτερ. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι ασχολούμαι με την υπόθεση αυτή με το Τατζικιστάν. Είμαι εισηγητής, ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την περιοχή εκεί οι 26 χώρες πρέπει να ξέρετε έχουν ήδη επικυρώσει τη συμφωνία και έτσι ελπίζουμε ότι και η Ελλάδα θα το κάνει το φθινόπωρο. Εξαρτάται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κατά πόσο τελικά θα δώσουμε την σύμφωνη γνώμη πριν από αυτή τη συμφωνία μετά. Έχουμε δύο κείμενα μπροστά μας. Έχουμε από την μια την πρόταση ψηφίσματος και από την άλλη το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Εξηγούμε ποια είναι τα προβλήματα στην ε, χώρα, λέμε τι συστάσεις κάνει η διεθνής κοινότητα προς το Τατζικιστάν για να δούμε πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση εκεί. Ελπίζω επίσης οι συνάδελφοι να βελτιώσουν την πρόταση αυτή ψηφίσματος μέχρι τις 25 Αυγούστου. Πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός και πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι στο Τατζικιστάν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα το πρόβλημα ένδυας με μια πολύ αδύναμη οικονομία οι φυσικοί πόροι είναι πολύ περιορισμένοι, δεν έχουν αποθέματα πετρολαίου ή φυσικού αερίου. Τελευταία βλέπουμε και τις συνέπειες από την οικονομική κρίση στην Ρωσία και στο Καζακστάν, όπου εργάζονται πολλοί ε, πολίτες του Τατζικιστάν και στέλνουν έτσι χρήματα στη χώρα τους. Στο Τατζικιστάν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, αλλά δεν υπάρχουν ε, συνθήκες δημοκρατικές με την έννοια που εμείς καταλαβαίνουμε αυτόν τον όρο. Πρόκειται για μια χώρα όπου υπάρχει μια κυβέρνηση ενός και μόνο κόμματος και στην έκθεση θα βρείτε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό η κοινωνία των πολιτών δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τα πράγματα. Επίσης έχουν ε, υιοθετηθεί πρόσφατα διάφοροι νόμοι στη χώρα που δυσκολεύουν πολύ την λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων εκεί. Επίσης έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις περιορισμού ελεύθερης ε, θρησκείας. Δηλαδή ο καθένας να, δεν μπορεί να έχει και να δράσει σύμφωνα με την θρησκεία του. Πάντως, η χώρα αυτή, το Τατζικιστάν, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην περιοχή. Υπάρχει δυνατότητα η χώρα αυτή να γίνει μια σύγχρονη χώρα. Μια χώρα που να μπορεί να ενισχύσει και τον ρόλο της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού, ε, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την ε, ανάπτυξη του Τατζικιστάν και να βελτιώσουμε τη, και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Θέλουμε επίσης να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία συνεργασίας και σύνδεσης. Τον Ιούνιο του 2007 υιοθετήσαμε τη στρατηγική μας για την Κεντρική Ασία. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ανέκρινε μια ειδική έκθεση του κυρίου Ιουτς όπου αναφέρεται ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν πέντε πολύ διαφορετικές μεταξύ τους χώρες, με εντελώς διαφορετικές συνθήκες και είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν καθορίζουμε τις πολιτικές μας. Χαίρομαι πάντως που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέκρινε τη θέση αυτή με την οποία συμφωνώ και εγώ. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να επιτρέψει να έχουμε μια αδύναμη χώρα και ασταθεί στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα προς το Τιτζικιστάν και να τους πούμε ότι είμαστε διατεθειμένοι για μια πιο στενή συνεργασία με αυτή τη χώρα. Πρέπει να προωθηθούν βέβαια εκεί οι μεταρρυθμίσεις που περιμένει ο κόσμος πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, πρόκειται για την καταπολέμηση της ένδυας ή για άλλα θέματα. Ελπίζουμε λοιπόν μέσω της στήριξής μας, της αρρωγής μας και του διαλόγου με τη χώρα αυτή να πετύχουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Το Τατζικιστάν από τη δικά του την πλευρά έχει πει ότι τη θέλει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές φορές το έχει πει, όπως επίσης θέλουν και εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πιο υψηλό επίπεδο. Θέλουν επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μας υπέρ της ανάπτυξης. Από τη δικιά μας την πλευρά θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα στο θέμα του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας, της εκπαίδευσης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και επίσης θέλουμε το Τατζικιστάν να πάρει στα σοβαρά τέτοιου είδους υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Εδώ πρέπει να πούμε επίσης ποια είναι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συμφωνία στο άρθρο 2 συγκεκριμένα, όπου λέει ότι η χώρα πρέπει να σεβαστεί τις αρχές της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα Και στην πρόταση ψηφίσματος ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της συνεργασίας με το Συμβούλιο να πετύχει πολύ στα σοβαρά να λυθούν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε επίπεδο, στο διάλογο δηλαδή που έχουμε με το Τατζικιστάν. Επίσης ζητάμε να στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Τατζικιστάν σε όλα τα επίπεδα που χρειάζεται. Κάνουμε επίσης έκκληση στους διεθνείς δωρητές προκειμένου αυτοί να προσανατολίσουν τα μέσα τους στην τοπική κυβέρνηση και στην κοινωνία των πολιτών του Τατζικιστάν με κάθε διαφάνεια. Τέλος, θέλω να προσθέσω πως πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να έχουμε μια πιο στενή συνεργασία με το Τατζικιστάν στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Συνεπώς, σας ζητώ να στηρίξετε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι πολύ καλή εργασία του συναδέλφου. Συμφωνούμε. Μας πράσινη, πράγματι είναι πολύ φτωχή χώρα το Τατζικιστάν. Θα έπρεπε ίσως να αναφέρουμε και την παιδική εργασία εδώ πέρα ως πρόβλημα. Αλλά το Τατζικιστάν έχει φυσικούς πόρους, υδροηλεκτρική ενέργεια π.χ. Και τυχαίνει να γνωρίζω πως η Κίνα σκοπεύει να κάνει μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Μιλάμε για 650 εκατομμύρια ευρώ θα ήθελα λοιπόν να καταθέσω μία τροπολογία για να παρακολουθήσουμε τις περιβαλλοντικές ε, συνέπειες ε, των ε, έργων αυτών για τα φράγματα. Είμαι σίγουρος πως είμαι σίγουρο πως έχει δίκιο ο εισηγητής, είναι διαφοροποιημένη στρατηγική μας εκεί πέρα στην ε, Κεντρική Ασία. Είναι σαφές πως το Τουρκμενιστάν είναι χειρότερο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Τατζικιστάν, αν και τα προβλήματα του Τατζικιστάν αναφέρονται πολύ καλά στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Τέλος, ως μέλος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κανονικά τα πράγματα αυτά τα εξετάζουμε εκ των προτέρων. αλλά τώρα ο χρόνος πιέζει, αλλά χαίρομαι που συμπεριέλαβε η εισηγητή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Γκάλερ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον συνάδελφο τον κύριο Πέτρελα για τις εξηγήσεις του. Κατά βάση, συμφωνώ με τα συμπεράσματα του σχέδιου ψηφίσματος, αν και ίσως εκεί που περιγράφεται η πολιτική κατάσταση θα έπρεπε να υπάρχει μια επικαιροποίηση. Δεν ξέρω από πότε είναι το κείμενο. να Έχει σημερινή ημερομηνία, αλλά οπωσδήποτε έχει γραφτεί παλιότερα. Το σημείο λέει στα αγγλικά αναγνωρίζει πως το Τατζικιστάν είναι σχετικά σταθερή χώρα χωρίς ενδείξεις εξωτερικής απειλής ή κάποιας εσωτερικής εξέγερσης κτλ. κτλ. Νομίζω την τελευταία εβδομάδα λάβαμε ενισχυτικές ειδήσει. Δηλαδή κάποιος υπεύθυνο για τον εμφύλιο προδεκαετίας ε, που είχε διαφύγει στο Αφγανιστάν ή Πακιστάν λόγω της αυξημένης πίεσης στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν με κάποιους δικούς του φαίνεται ότι επανήλθε στη χώρα και είναι σύμμαχος των Ταλιμπάν αυτός. Οπότε ο νότος της χώρας από ό,τι φαίνεται αποτελεί πεδίο δράσης αυτών των ανθρώπων. Οπότε όταν μιλάμε για σταθερή χώρα πρέπει να το επικαιροποιήσουμε αυτό. Έχουμε συγκεκριμένο κίνδυνο ε, αποσταθεροποίησης μέσω αυτών των δυνάμεων. Ακριβώς γιατί η κυβέρνηση εν ενεργεία δεν είναι και ιδιαίτερα έτσι δημοκρατική ή επιτυχής στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα και δεν βρίσκει άρα και μεγάλη στήριξη. Θεωρώ πως τελικά πρέπει να κλείσουμε τη συμφωνία γιατί έχουμε συμφέρον να σταθεροποιηθεί η χώρα, μην έχουμε ψευδεστήσεις ως επικρατεί όμως καμία κατάσταση που μπορεί να περιγραφεί και ως σταθερή. Ευχαριστώ. Intervento l'onorevole e passo la Ευχαριστούμε τον Αφρικάρη και το λόγο στον Σαν Φαρλάκη. Συμφωνώ με το κείμενο, με την εισηγήτρια. ως θεμαρχής. Θα προτιμούσα όμως μια πιο ενδελεχή αναφορά στο Τζικιστάνο χώρα από το, που, το οποίο περνάει το μεγαλύτερο τμήμα της ε, αφγανικής ηρωίνης προς τη Ρωσία και την Ένωση. Γι' αυτό η χώρα είναι σημαντική για μας και γι' αυτό υπάρχουν σοβαρές, τόσο σοβαρές παραβάσεις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέρασε από ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο με 150.000 και νεκρούς το 1997 τελείωσε και η σταθεροποίηση της χώρας εν μέρη οφείλεται στο ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των κύριων πολιτικών και εγκληματικών οργανώσεων της χώρας. Στο Τατζικιστάν ο πόλεμος ουσιαστικά ήταν πόλεμος μεταξύ διαφόρων συνασπισμών ομάδων και ήταν και το αντικείμενο παρέμβασης των Ηνωμένων Εθνών και όσον αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης με επιτυχία, παραμένει επιτυχής η παρέμβαση αυτή, το Ηνωμένο, ε, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ένα, μια ε, ε, αποστολή η οποία προσπάθησε να εμποδίσει την ροή αυτή ηρωίνη προς τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη. Η υπηρεσία αυτή των ΗΕ κατάσχεσε πάνω από τρει τόνους ηρωίνη σε λίγα χρόνια και ουσιαστικά χρηματοδοτείται από την Ένωση. Το κείμενο είναι σωστό όσον αφορά την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και όσον αφορά τις προτάσεις. Εγώ όμως θα ήθελα να τονιστεί περισσότερο ποια είναι η κύρια αιτία της φτώχειας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χώρα είναι πανφτωχή. Ο ένας στους δύο είναι κάτω από τη γραμμή της φτώχειας. Είναι από τις πιο φτωχές χώρες μεταξύ των πέντε δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας και θα ήθελα αυτό να τονιστεί τα χρήματα της Ένωσης θα πρέπει να πάνε άμεσα σε πρωτοβουλίες μείωσης στις στόχης. Διαφορετικά θα εξακολουθήσουμε να είμαστε μάρτυρες αυτών των σοβαρών παραβιάσεων. Γιατί είναι κληρονομιά και του εμφύλιου πόλεμου και της σύγκρουσης μεταξύ του Ισλαμισμού και άλλων δυνάμεων Δεν ξέρω αν θα κάνω τροπολογία, γιατί δεν το σκέφτηκα μέχρι τώρα το θέμα αυτό ως τροπολογία. Πάντως, ε, προτείνω να υπογραμμιστεί το σημείο αυτό πολύ πολύ περισσότερο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον κύριο Αρλάκη. Δεν ζήτησε κανένας άλλος συνάδελφο το λόγο. Το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, κύριος Μπέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, συγχαίρω το εισηγητή κύριο Πέτερλε για το εντολή που του δόθηκε. Άκουσα με προσοχή την ανάλυση του και τις ε, ερωτήσεις που ετέθησαν από τους ε, ευρωβουλευτές. κατάσταση είναι δύσκολη. Γιατί έχουμε ειδήσει σχετικά με θέματα εσωτερικής ασφάλειας και είναι νωρίς να πούμε που θα καταλήξει αυτή η κατάσταση, πάντως μας ανησυχεί. Το Τατζικιστάν παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την μείωση της βίας και του εξτρεμισμού από τη μεριά του Αφγανιστάν. 1.300 χιλιόμετρα κοινά σύνορα έχει με το Αφγανιστάν και θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές για συγκεκριμένα προγράμματα και όσον αφορά τη μακροασφάλεια, γιατί υπάρχει κίνδυνος να έχουμε ε, εξτρεμισμό ισλαμικού χαρακτήρα από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν να επεκταθεί και προς άλλες κατευθύνσεις, αλλά και για λόγους μικροασφάλειας, όπου η καταπολέμηση λαθρεμπορίων ναρκωτικών και οργανωμένου εγκλήματος γενικά. Στην επίσκεψη του Πρόεδρου του Τατζικιστάν του Φεβράριο στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος Μπαρόσο εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την ασφάλεια της περιοχής λόγω της ασταθούς κατάστασης στο Αφγανιστάν. Στη χώρα υπάρχει ένα πρόβλημα λόγω του ότι είναι ασθενές κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα και δεινά της χώρας. Η ενεργειακή υποδομή είναι ανεπαρκής. Προκειμένου να έχει ηλεκτρισμό όλη η χώρα τα εμβάσματα των μεταναστών που ήταν ο κινητήρας της οικονομίας έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έχουν μειωθεί κατά 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια και αν συνεχιστεί αυτό και τον επόμενο χειμώνα η Κομισιόν ανησυχεί για τον κίνδυνο κοινωνικής αναταραχής και πολλοί μετανάστες μπορεί να επιστρέψουν από τη Ρωσία στη χώρα λόγω τη οικονομική κρίση ιδιαίτερα στις οικοδομές στη Ρωσία. Πολλοί Τατζίκοι δουλεύουν στη Ρωσία και θα επιστρέψουν. Μα ανησυχεί αυτό. Η χώρα είναι, έχει ρόλο κλειδί στην εφαρμογή τη πολιτική μα για την Κεντρική Ασία τη σταθεροποίηση, όπω αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007. Θέλουμε να έχουμε περισσότερη συνεργασία με τη χώρα αυτή από τη στιγμή που η εταιρική συμφωνία θα επικυρωθεί η Ελλάδα είπε ότι θα επικυρώσει τη συμφωνία το Σεπτέμβριο. Με αυτή την επικύρωση και με την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου θα ωφεληθούν οι σχέσεις μας με το Τατζικιστάν. Γιατί όπως σας είπα, η χώρα αυτή της Κεντρικής Ασίας είναι σημαντική για τη στρατηγική μας, για την περιοχή αυτή. Θα συνεργαστούμε με τη γραμματεία του Κοινοβουλίου να επικαιροποιηθεί το κείμενο. Μπορούσαμε να κάνουμε και ορισμένε μικροπροσθήκες, αν θέλετε, εγκαίρως πριν από την επόμενη συνεδρίασή σας του Σεπτεμβρίου ή και μετά στο Στρασβούργο. Τώρα για το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να καθησυχάσω τους ευρωβουλευτές ότι και αυτό μας, προ... προβληματίζει και μας. Ο πρώτος διάλογος ξεκίνησε τον Οκτώβριο πέρυσι. Υπάρχουν ορισμένα λεπτά θέματα, όχι ελευθερία μέσων ενημέρωσης. Στου στους κρατούμενους και φυλακισμένους. Η παιδική εργασία θεωρητικά είναι εκτός νόμου, αλλά έχουμε λοιπόν αυτό το διάλογο. Αυτό είναι θετικό πολιτικό σινιάλο και είναι απλώς μια αρχή. Πρόσφατα είχαμε ένα σεμινάριο σχετικά με την κοινωνία των πολιτών, επιτυχές, συμπλήρωσε το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέμα ήταν το δικαίωμα για μια, σε μια δίκαιη δίκη και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Είχαμε πολλούς εκπροσώπους και από Υπουργεία και από τις αρχές, ο διαμεσολαβητής, υπήρξε ένας κατάλογος συστάσεων Τέλος Αυγούστου θα οριστικοποιηθούν τα πορίσματα του σεμιναριού. Όντως το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα πρωτεύον θέμα, στοιχείο του πολιτικού διαλόγου, προβληματίζει και ενδιαφέρει την Κομισιόν επικροτούμε όλα όσα υπόθηκαν από τη μεριά του εισηγητή σήμερα. Και θα περιμένουμε και εμείς με ελπίδα την επικύρωση της συμφωνίας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μπέρν. Το λόγο για να κλείνουμε στον εισηγητή μας, τον κύριο Πέτερλε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ναι, δεν είναι πάντα βαρετό το τελευταίο ζήτημα της ημερήσιας διάταξης όπως έδειξε και η συζήτησή μας. Εγώ χαίρομαι γενικά και για την στήριξή σας. Σας ευχαριστώ για όλα τα σημεία τα οποία αναφέρατε, τις προτάσεις τις οποίες κάνατε και με τη βοήθειά σας θα προσπαθήσω να επικαιροποιήσω την έκθεσή μου. Πράγματι η έκθεση αυτή πέρασε μια ολόκληρη διαδικασία, δεν εγκρίθηκε στην προηγούμενη θητεία και τώρα ξανά ε, υποβάλλεται στην αρχή της νέας ε, θητείας. Οπότε πράγματι δικαιολογημένα μιλήσατε για επικαιροποίηση. Αναμένω λοιπόν μέχρι τις 25 Αυγούστου τροπολογίες και είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ μαζί σας και με την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Bene, ehm, Στο σημείο αυτό λοιπόν το μόνο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για τις τελευταίες διευκρινήσεις που μας έδωσε να του πω ότι εδώ βέβαια περιοριζόμαστε κάπως γιατί το Συμβούλιο ζήτησε το κατεπήγον για τη συμφωνία αυτή. Γιατί η διαδικασία επικύρωσης έχει προχωρήσει και είναι στο τελευταίο στάδιο. Συνεπώς έχουμε χρονικούς περιορισμούς. Αρχές Αυγούστου πρέπει να έχουμε τις τροπολογίες για να μπορέσουμε μετά στην Επιτροπή μας να εγκρίνουμε τις τροπολογίες αυτές. Βέβαια υπάρχει και άλλο προηγούμενο, πάντως τις τροπολογίες μπορεί να μην τι έχουμε σε όλες τις γλώσσες, στα αγγλικά όμως θα τις έχουμε βέβαια. Ζήτησα την άποψή σας. Αν συμφωνούμε επί της ουσίας για την έγκριση της συμφωνίας αυτής, ε, νομίζω ότι έτσι καλώς όλοι να γνωρίζουμε πως είναι αποδεκτό πως τη χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία και τη σταθερότητα κτλ. Λοιπόν, ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίασή μας νομίζω. 1 ε, και 2 Σεπτεμβρίου συνεδριάζουμε και πάλι. Θα έχουμε τον Επίτροπο Λιρέν, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στα Βαλκάνια και την Τουρκία. Και μετά κρόση θα έχουμε με τον νέο αντιπρόσωπο του ΙΕ για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλές και ήρεμες διακοπές. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. <laughs>